Το ψήφισμα που θα εκδοθεί από το Κοινοβούλιο για όλα αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρος και εμείς ευχαριστούμε κύριε Βάμεν. Κλείνει λοιπόν η συζήτηση και θα ακολουθήσουν κάποιες ανακοινώσεις. Οι αρμόδιες αρχές της Πολωνίας κατέθεσαν αίτημα ε, για άρση της ασυλίας ε, του κυρίου Βαλένσα. Το αίτημα υποβλήθηκε στον πρόεδρο ε, και σύμφωνα με το καταστικό μας το αίτημα αυτό θα παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή από, την, από τους Σοσιαλδημοκράτες και την ΓΚΟΕ πήραν αίτημα για ορισμούς ε, αρμοδίων και μελών σε επιτροπές. Ε, έχει συμπεριληφθούν αυτοί οι ορισμοί στα πρακτικά. Ε, μέχρι να εγκρινθούν τα πρακτικά μπορείτε να προσθέσετε να κάνετε αλλαγές σε αυτούς τους ορισμούς μελών. Πάμε στην έκθεση Γκεμπράντι και θα ήθελα καταρχήν να δώσω το λόγο στον κύριο Γκεμπράντι για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ξεκινήσω με κάποιους ε, αριθμούς ε, ε, που πολλοί μόνο τους φανταστούν μπορούν, άλλοι πάλι όχι. Δηλαδή το 2050 θα είμαστε εννέα δις άνθρωποι σε αυτή τη γη και μέχρι τότε θα έχουμε διπλασιασμό της μεσαίας τάξης με μέσο εισόδημα ε, μέχρι 3 δις ε, και τώρα ε, έχουμε καταναλώσει ήδη δύο πλανήτες. Μέχρι τότε θα χρειαστούμε τρεις πλανήτες που δεν θα υπάρχουν. Η δική μας λοιπόν η οικονομία διψάει για φτηνούς πόρους, ε, μειώνονται οι φτηνοί πόροι και αυτό κοστίζει ε, στις χώρες μας δισεκατομμύρια. Άρα δηλαδή αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δράση για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Ο χάρτης ε, πορείας της Επιτροπής, συγχαίρω τον Επίτροπο, είναι μια πολύ καλή τάξη προς τη σωστή κατεύθυνση. Η ανάλυση και η προσέγγιση τη Κομισιόν είναι πάρα πολύ καλέ. Αυτό που κατά την άποψή μου λείπει είναι ότι δεν υπάρχει η κατεπίγουσα μορφή σε αυτή την έκθεση. Ακριβώ λοιπόν αυτό θέλουμε να καταστήσουμε σαφέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται μόνο για το περιεχόμενο τη έκθεση, αλλά πρόκειται και για τη δομή τη, όπου ε, στην Επιτροπή περιβάλλοντο, εμεί εντοπίσαμε έξι ε, ουσιαστικά σημεία. Τα αναφέρω ε, με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα είναι ιδιαίτερα σημαντικό από κοινού με τις επιχειρήσεις να ε, εκπονήσουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης έτσι ώστε στις επιχειρήσεις της Ευρώπης να επικρατήσει αποτελεσματικότερη χρήση των φυσικών πόρων. Για να γίνει αυτό οι εταιρείε, οι επιχειρήσεις πρέπει να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο έτσι ώστε να έχουν ε, παραγωγή, εκμετάλλευση πόρων με ε, κάποια συνειδητοποίηση. Χρειαζόμαστε και την ανακύκλωση. Ε, θα πρέπει να είναι ευκολότερο πρώτες ύλες ε, να τις κυκλοφορούμε και ανακυκλώνουμε και εδώ εντάσσονται και οι δευτερογενείς ε, πρώτες ύλες που χρειάζονται δημοσιονομική ενίσχυση για να καταστούν αυτές φτηνότερες από τις πρώτες ύλες. Ε, έρευνα και ανάπτυξη. Πρέπει να αναπτύξουμε εκεί εναλλακτικέ λύσεις, να στηρίξουμε τον τομέα της ανακύκλωσης, να γίνει αυτός πιο επαγγελματικός. Τέταρτον, οφείλουμε να επεκτείνουμε τον οικολογικό σχεδιασμό. Μέχρι τώρα ισχύει μόνο για την ενέργεια, αλλά θέλουμε να αποδείξουμε ότι και οι πρώτες ύλες μπορούν να ανακτηθούν. Όλα αυτά ξεκινάνε στη φάση του σχεδιασμού. Κατόπιν, οφείλουμε ε, να εξετάσουμε ε, ή το θέμα της ε, οικονομικής μεταχείρισης των πόρων πρέπει να τον επεκτείνουμε και σε άλλους τομείς όπως τη γεωργία ή στην αλία και η έκτη σημαντική προτεραιότητα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν σε ολόκληρη την Ευρώπη σαφείς δείκτες με βάση την άποψη του Κοινοβουλίου θα πρέπει να επεκταθεί το αποτύπωμα. Είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Πρόεδρε, έχω δουλέψει πάρα πολύ για όλα αυτά τα θέματα και έχω πλέον ε, παρατηρήσει ότι εδώ δεν πρόκειται για οικολογικό αλλά για οικονομικό πρόβλημα. Οφείλουμε να μεριμνήσουμε έτσι ώστε όλα αυτά μακροπρόθεσμα να είναι πιο οικονομικά. Ανέφερα ότι οι επιχειρήσεις ε, χρειάζονται περισσότερα δισεκατομμύρια για τις πρώτες ύλες διότι αυξάνονται οι ε, τιμές των πρώτων υλών. Περί αυτού πρόκειται. Και δυστυχώς το Συμβούλιο σήμερα δεν είναι παρόν. Λυπάμαι πάρα πολύ που το Συμβούλιο δεν μοιάζει να ενδιαφέρεται ε, για να επιτευχθούν περισσότερα στην Ευρώπη και να ακολουθήσουμε ένα καλύτερο δρόμο απέναντι στη μεταχείριση των πρώτων υλών. Ο κ. Ποτότσνικ εκ μέρους Επιτροπής έχει το λόγο. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώτα θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Γκυμπράντη για την έκθεσή του που αναγνωρίζει το, ένα υψηλό βαθμό αισιοδοξία που απαιτείται για την ε, δημιουργία μια ασφαλού Ευρώπη. Αναφέρεται και στην πολιτική σημασία του, της επάρκειας και τις ανάγκες να ληφθούν μέτρα ώστε να ανταποκριθούμε στις οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Οι περιορισμοί των πόρων είναι μια τάση διεθνής την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η οικονομική κρίση έχει αποδείξει την ανάγκη για επίγουσες ανάγκες σε επίπεδο οικονομία και την ανάγκη επίση να εξετάσουμε καλύτερα το αναπτυξιακό μας μοντέλο. Χωρίς νέες πολιτικές θα ασκηθούν μεγαλύτερες πιέσεις στο περιβάλλον και δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε τους στόχους μας για την κλιματική αλλαγή και θα εκθέσουμε την οικονομία και την ευημερία μας σε συστημικούς κινδύνους η, βιώσιμη χρήση των πόρων είναι η προϋπόθεση για μακροχρόνια ε, ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα των οικονομιών μας. Αυτή είναι επίσης και μια πολλά υποσχόμενη πηγή για θέσεις απασχόλησης και ευκαιρίες για τους ε, ε, επιχειρηματίες βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Η Επιτροπή έχει παρουσιάσει το όραμα της στα πλαίσια της μακροχρόνιας στρατηγικής με την ε, πρωτοβουλία 2020 που καλύπτει την ενέργεια, το νερό, την βιοπικιλότητα, τις μεταφορές κλπ. Έχουμε εντάξει την αποτελεσματικότητα αυτή στις προσπάθειές μας για συνοχή, για τη γεωργία, για την και κλπ. Και ελπίζω ότι τα αποτελέσματα της νομοθετικής διαδικασίας θα είναι αντάξεις των φιλοδοξιών μας ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος μέσα από αυτό το πρόγραμμα έχουμε θέσει στο τραπέζι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για να τηρήσουμε τον ε, στόχο της βιωσιμότητας το 2020. Έχουμε προβλέψει μια διαδικασία που θα θέσει σε κίνηση αυτή τη διαδικασία. Αντιμετωπίζουμε τα θέματα από τρεις ε, οπτικές γωνίες και με τα χαράς βλέπω ότι συμμερίζεται την άποψή μα προ τι προτεραιότητε στην έκθεσή σας. Πρώτον, υπογραμμίζουμε την ανάγκη να εξασφαλίσουμε τι οριζόντιε συνθήκε για την μετάβαση τη οικονομία. Εξετάζουμε την κατανάλωση και την παραγωγή και ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και υπογραμμίζουμε την ανάγκη για την έρευνα και την καινοτομία και τη σημαντική ανάγκη να διακόψουμε τις ε, ανεπαρκείς, ε, τις ε, μη αποτελεσματικές επιδοτήσεις. Είναι σημαντικό να ενισχύσουμε την παραγωγικότητα της οικονομίας και της ανάπτυξης. Η πλήρης εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας θα μας επιτρέψει να οικονομήσουμε 70 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Να αυξήσουμε την ετήσιο τζίρο κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων και να δημιουργήσουμε πάνω από 400.000 θέσεις εργασίας μέχρι το 2020. Δεύτερον, η φύση του στόχου που επιδιώκουμε. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το φυσικό μας κεφάλαιο και τα οικολογικά συστήματα που προσφέρει θα ισχύουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα γιατί είναι το εχέγγυο για την ποιότητα ζωής μας υπάρχουν πόροι τους οποίους προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπάρχουν τομείς που θεωρούμε ότι είναι οι πιο σημαντικοί ε, για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ε, τα τρόφιμα, οι μετακινήσεις και οι μεταφορές και με τα χαράς βλέπω ότι αυτό είναι και στην έκθεσή σας μια σταθερότητα. Η απόδοση των πόρων σημαίνει ένα πρόγραμμα ένταξης και ενσωμάτωσης και εσείς είστε αποφασισμένοι να επιφέρετε τις αναγκαίες αλλαγές. Στη διάρκεια του εξαμήνου θα εξασφαλίσουμε ότι ακολουθούν τη σωστή πορεία όλα τα κράτη-μέλη. Θα κινήσουμε μια διαδικασία για να προσδιορίσουμε τους στόχους που απαιτούνται για αποτελεσματικούς δείκτες που να βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα μέχρι το 2013. Φυσικά χρειαζόμαστε επίσης απόλυτη εφαρμογή Τη περιβαλλοντική νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με δράση σε εθνικό επίπεδο ώστε να εξασφαλίσουμε ίσου κανόνε για όλου. Όπω πάντα, οι δεσμεύσει όλων των ενδιαφερομένων μερών είναι σημαντικέ για την εφαρμογή του προγράμματο. Πρέπει να κινητοποιήσουμε του παίκτε σε όλα τα επίπεδα και σε όλου του σχετικού τομεί, ώστε να αναλάβουν και εκείνοι τι ευθύνε του. Υπολογίζω στην υποστήριξή σα. γι' αυτό. Θα παρακολουθήσω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την σημερινή συζήτηση και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Επιτροπέ Ποτότσνικ. Τώρα, ο κύριος Γιακολίνο, δύο λεπτά από την ΙΝΤΑ, ε, από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μόλις άκουσα τον κύριο Κερμπράντη και άκουσα και τον Επίτροπο Ποτόσνικ. Είμαι ο εισηγητής της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Σημειώνω θετικά ε, ότι ε, το κείμενο αυτό της Επιτροπής Περιβάλλοντος ε, συμπεριλαμβάνει πάρα πολλές παρατηρήσεις που έχουμε κάνει σχετικά με το διεθνές εμπόριο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ε, στο εξωτερικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το εμπόριο αγαθών είναι ένα εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης πάρα πολύ σημαντικό. Κυρίως το άνοιγμα των αγορών για αγαθά και υπηρεσίες και η ε, κατανάλωση ενέργειας που σχετίζεται με αυτά τα αγατά ε, μπορούν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας ε, και νέες να προάγουν τις νέες τεχνολογίες. Ε, η ανταγωνιστικότητα ξεκινάει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εμείς λοιπόν στη γνωμοδότηση επιβεβαιώνουμε ότι ορισμένα σημεία είναι πολύ σημαντικά στις ε, διμερείς και πολυμερείς αλλά και περιφερειακές συμφωνίες που συνάπτονται ο περιορισμός των δασμολογικών και μη δασμολογικών εμποδίων, η ανταλλαγή προϊόντων, η συμπερίληψη ενός κεφαλαίου ε, σχετικά με την βιωσιμότητα. Ε, αυτά είναι πολύ σημαντικά για ό,τι παράγεται στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων. Είναι σημαντικό να απλουστευτούν οι διαδικασίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να παραμείνει ηγέτιδα δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο και να προάγει με το εμπόριο, αγαθά ε, και ε, πράσινες υπηρεσίες οφείλουμε να ασκήσουμε πίεση κυρίως απέναντι σε τρίτες χώρες για εμπορικές ε, συμφωνίες που θα είναι συνεπείς με μέτρα ενεργειακής απόδοσης έτσι ώστε κύριε Πρόεδρε να έχουμε μια ουσιαστική και ευφυή ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε κύριε Γιακολίνο, εκ μέρου τη Επιτροπής ε, Βιομηχανίας, Συνάδελφο κύριο Γιώχανσον για ένα λεπτά. Ένα λεπτό, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, η, ο εισηγητή μα ε, μας παρουσίασε την έκθεση. Εγώ είμαι η εισηγητή τη Επιτροπής Βιομηχανίας για το θέμα αυτό και θα ήθελα να πω ότι δεν έχουμε αντίφαση στην πρόταση αυτή, αλλά μία υπόσχεση για καλύτερη ανταγωνιστικότητα στην ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε καινοτόμα ευρηματικά επιχειρηματικά μοντέλα, έρευνα, καινοτομία, καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας για το οικολογικό design και την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα. Στην γνωμοδότηση της ΙΤΡΕ ασχολούμαστε και με ένα άλλο θέμα. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους ε, ώστε οι βέλτιστες πρακτικές των κρατών μερών εφαρμοστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, να έχουμε δείκτες, ποσοτικοποιημένους στόχους, συγκεκριμένο τρόπο για να αποτιμήσουμε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες. Χρειαζόμαστε και μηχανισμούς φυσικά χρηματοδότησης ε, των διαφόρων προτάσεων. Όλα αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά και για την αξιοποίηση των πόρων μας. Αγαπητούμε, ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρους της ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης, ο συνάδελφος κ. Βον για ένα λεπτό. Uh, uh, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, με ιδιαίτερη ικανοποίηση συνέταξε γνωμοδότηση για την ε, έκθεση αυτή και Χαιρόμαστε για το ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι ευληματική πρωτοβουλία του 2020. Επίσης, ζητούμε περισσότερες επενδύσεις στις υποδομές για σχέδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και χαίρομαι ότι ο νέος ε, κανονισμός για την πολιτική συνοχή συλλαμβάνει και αυτό το θέμα υπόψη. Επίσης ζητήσαμε ενίσχυση της ε, συμβολής ε, συνεισφοράς των διαρθρωτικών ταμείων για προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης. Και φυσικά η πολιτική συνοχή το λαμβάνει και αυτό υπόψη. Ζητήσαμε και ενισχυμένο συντονισμό μεταξύ των διαφόρων κοινοτικών ταμείων, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τέτοια ενεργειακή απόδοση. Γι' αυτό και προτείνουμε εναρμόνιση των διαρθρωτικών ταμείων στο μέλλον. Η Επιτροπή μα ε, ζήτησε καλύτερο συντονισμό μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Γιατί σε τελική ανάλυση τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ ε, είναι αυτέ ε, που θα εφαρμόσουν εμπράκτω αυτά τα σχέδια και προγράμματα. Αν κατακλείδη λοιπόν η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι ικανοποιημένη με την έκθεση της κατουσίαν αρμόδιας Επιτροπής. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθούν τώρα εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Ε, καταρχήν ο συνάδελφος κ. Φλόρεντς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Ποτότσνικ. Σας συγχαίρουμε θερμά για αυτή την ε, θαραλέα έκθεση η οποία δεν είναι απλά μια έκθεση περί πόρων που στον εμπλουτισμό της ζωής μας. Κοιτάξτε, η ε, επάρκεια πόρων δεν είναι κάτι που ε, ευαγγελίζονται οι θεροβάμονες είναι μια πραγματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να εξετάζουμε το θέμα και από το, κάτω από το πρίσμα της ανταγωνιστικότητας. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να γίνεται αυτή η συζήτηση χωρίς ε, την ίδια στιγμή να ζητάμε νομοθεσία. Υπάρχουν πολλοί κανόνες. Με κανόνες μπορούμε να λύσουμε το θέμα, να επισημάνουμε στη βιομηχανία πόσο αποτελεσματικότεροι μπορούμε να γίνουμε.

Ε, ο πατέρας μου το προσπάθησε, εγώ το προσπάθησα με τα παιδιά μου. Ε, κοιτάξτε, ο δρόμος που έχουμε ακολουθήσει μέχρι τώρα δεν είναι αποτελεσματικός. Πρέπει να βρούμε ένα δρόμο αποτελεσματικότητα. Είχα ένα αυτοκίνητο με 12 λίτρα, ε, τώρα έχω ένα με 7 και θα πάμε στα 3. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Και τι ήταν λάθος αυτό που οι γονείς μας μας έλεγαν, ότι η αποτελεσματικότητα είναι αυτό που γίνεται με το δάσος. Ε, δηλαδή να παίρνει κανείς από το δάσος μόνο τόσα ξύλα όσα θα αναπτυχθούν στη διάρκεια ενός έτους. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστώ θερμά τον συνάδελφο κύριο Γκεμπράντι που είναι πάρα πολύ ευχάριστο να συνεργάζεται κανείς μαζί του. Ε, θέσαμε σωστά θεμέλια. Βεβαίως από τους πολιτικούς μου φίλους από την άλλη πλευρά υπάρχουν υπερβολές. Πραγματικά θέλετε να απαγορεύσετε την κατανάλωση κρέατος. Πραγματικά λέτε ότι σε κάθε κάθε λογαριασμό θα πρέπει να αναφέρεται ποιο είναι το οικολογικό αποτύπωμα. Και ε, κάποιο ε, που δεν θα το τηρεί αυτό, ε, τι θα γίνεται με αυτόν, σα παρακαλώ πάρα πολύ, α μην τα λέμε αυτά. Κατόπιν, η προσέγγιση με του συντελεστέ είναι σωστή, αλλά και αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να ελοπιθεί εν μια ανοιχτή. Στην Συνάδελφε κύριε Γκεμπράντι, θα προσπιθεί προσπαθήσουμε από κοινού να διαγράψουμε τις ανοησίε και να προβάλλουμε τα σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, ε, συνάδελφε Φλόρεντ, η κυρία Μέρκη ακολουθεί. Ευχαριστώ κύριε, Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, έσπασε ο βραστήρας μου και δεν μπόρεσα να τον διορθώσω, να τον επισκευάσω. Διότι είμαστε, ζούμε σε μια κοινωνία που προτιμάμε να αγοράζουμε ένα νέο προϊόν παρά να επισκευάσουμε ένα παλιό, γιατί αυτό κοστίζει ακριβότερα. Πρέπει να θέσουμε τέρμα σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να μιλήσουμε για τη, τους πόρους το 2007 είχαμε την έκθεση της Λέσχης της Ρώμης που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Έχουμε φτάσει τώρα στο 2012 και δεν έχει λυθεί το θέμα, ούτε και τα επόμενα 40 χρόνια θα λυθεί. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι, το συγκεκριμένο μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν δύο στρατηγικέ που μας παρουσιάστηκαν για τις πρώτε και τώρα έχουμε την απόδοση και την αποτελεσματικότητα των πόρων. Όλα αυτά πρέπει να ενταχθούν στις κοινωνίες μας με έναν τρόπο ο οποίος θα επιτρέψει στους νέους να μην ε, υπερκαταναλώνουν, να μην, να, ώστε να, υπάρξει, να υπάρξουν οι πόροι να είναι διαθέσιμοι για όλους. Έχουμε πρόταση για ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο που δεν μιλάει για αντικατάσταση αλλά για επισκευή. Χρειαζόμαστε νέα μοντέλα και όχι νέες τεχνολογίες. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να τονίσουμε. Καλύτερη επισήμανση των προϊόντων, μία για την ενεργειακή απόδοση, μία για, για άλλα πράγματα, πέντε συνολικά ετικέτες, να οργανώσουμε καλύτερα τα συστήματα ανακύκλωσης, αποφεύγοντας την αποτέφρωση ε, ε, γιατί χρησιμοποιούμε τρία ε, γήπεδα ποδοσφαίρου. Αυτό ε, επιβαρύνει το περιβάλλον. Αρκεί ένα γήπεδο ποδοσφαίρου για την ενέργεια και για την διατροφή μας. Και κάτι ακόμα, το 2006 χρειαζόμαστε 200 δολάρια. Τώρα χρειαζόμαστε 600 το ποσό πολλαπλασιάστηκε σημαντικά σε τρία χρόνια. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε το συντομότερο για να διασώσουμε την οικονομία μας και το περιβάλλον μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ο συνάδελφος Παναγιώτοφ για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η παρούσα κρίση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αντιμετωπίζει υψηλή ανεργία, οικονομική ύφεση, Προκλήσει που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε άμεσα. Υπάρχουν όμω και άλλα προβλήματα που δεν φαίνονται εκ πρώτη όψεω και επίση χρήζουν άμεση ε, επίλυση, Όπω ε, το θέμα τη ε, αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. θα αυξηθεί ραγδαίο ο παγκόσμιο πληθυσμό τα επόμενα χρόνια και θα πρέπει και οι αναπτυσσόμενε χώρε να δρέψουν τους καρπούς της εργασίας τους στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Να μην ξεχνάμε όμως ότι οι παγκόσμιοι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα όρια τους και να αλλάξουμε τις συνήθειές μας για υπερβολική κατανάλωση πόρων. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε βιώσιμη και αηφόρα ανάπτυξη. Επίσης θα πρέπει να έχουμε και εναλλακτικό καινοτόμο πρόγραμμα που θα δίνει έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση των πόρων και στην καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αν θέλουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα της ε, ασφάλειας των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποφύγουμε σπάνι ε, και ανεπάρκεια, γιατί οι πόροι εξαντλούνται παγκοσμίω. Τα παγκόσμια προβλήματα χρήζουν παγκόσμια ε, λύσης. Δεν θα πρέπει να μείνουμε απογορωμένοι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πρωτοστατήσει διεθνώς και να βελτιώσει το πρόγραμμά της για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Ευχαριστώ θερμά τον συνάδελφο για την καταπληκτική του έκθεση και τον κύριο Επιτροπό για την παρουσίαση που μας έκανε. Ευχαριστούμε κύριε Παναγιώτοφ, ο κύριος Χόουτ για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή μας για την έκθεση που εκπώνησε εμένα μου τράβηξαν την προσοχή οι αιτήσει εκθέσει των μεγάλων επιχειρήσεων, των πολυεθνικών. Η Άξο Νόμπελ, για παράδειγμα, αναφέρει ότι η αυξήσει τιμών των ε, βασικών πόρων είχε ως συνέπεια για την εταιρεία ε, περιορισμό, σημαντικό περιορισμό του περιθωρίου κέρδους. Αναφέρεται στην ετήσια έκθεση ότι η εταιρεία αυτή πραγματοποιεί λιγότερα κέρδη λόγω της αύξησης των τιμών. Και δεν μπορούν να μετακυλήσουν αυτή την αύξηση των τιμών ε, στους καταναλωτές. Το ίδιο ισχυρίζεται και η Unilever. Λέει ότι πλήρωσε 2,5 δισεκατομμύρια τον περασμένο χρόνο. Μια πολυεθνική λοιπόν που επίσης λέει ότι η αυξήσει των τιμών ε, των, ε, των πρώτων υλών έχει επίδραση στη, στο κέρδος. Μιλάμε για ένα θέμα που αφορά την οικονομία και όχι μόνο τους πράσινους. Όλες οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για κάτι τέτοιο. Στις κάτω μόνο μία στι μόνο μία στι πέντε επιχειρήσεις έχει μία στρατηγική αντίθραση απέναντι στις αυξήσεις των τιμών των πρώτων υλών. Μόνο μία στις πέντε εταιρειε έχει τέτοια στρατηγική. Ενώ θα πρέπει όλοι από κοινού να ενδιαφερθούμε για την καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων και των πρώτων υλών μας. Έχουν ε, υποβληθεί πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, πολύ χρήσιμες, για παράδειγμα πώς θα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους σπόρους μας, πώς θα τους εξοπλίσουμε. Μπορούμε επίσης να ενδιαφερθούμε για το φορολογικό θέμα, ε, να εξασφαλίσουμε συμμόρφωση με τους ε, υπάρχοντες κανόνες για την ανακύκλωση για παράδειγμα ή για τα απόβλητα, να κάνουμε μια αναθεώρηση μεταρρύθμιση της ε, γεωργικής πολιτικής και να εκπονήσουμε και κάποιους δείκτες. Έχουμε μια πολύ καλή θεματολογία και πολύ χρήσιμες προτάσεις. Τώρα θα πρέπει να περάσουμε από τα λόγια στα έργα. Μια αποτελεσματική, αποδοτική και πράσινη οικονομία θα μα δείξει το δρόμο διεξόδου από την κρίση. Αλλά θα πρέπει να είμαστε σοβαροί στη δεσμευσή μα τι γίνεται με τα απόβλητα, τι γίνεται με τα γεωργικά απόβλητα, πώς θα χρησιμοποιήσουμε με υπεύθυνο και αποτελεσματικό τρόπο τις, ε, τα λοιπάσματα που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να μας ε, τραβήξουν την προσοχή για να φτάσουμε σε μια πραγματική οικολογική πράσινη οικονομία που είναι και η οικονομία του μέλλοντος για την Ευρώπη. Το λόγο κύριος Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, επιτρέψτε μου λοιπόν και εγώ να συγχαρώ τον συνάδελφο Γκεμπράντι για την έκθεσή του. Η φιντολή χρήση ε, των πόρων και της ε, παραγωγής είναι ένας ε, στόχος για όλους μας. Όμως στην έκθεση υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία για μένα είναι σχεδόν απαράδεκτα. Δεν λέω παντελώς απαράδεκτα, λέω σχεδόν απαράδεκτα, διότι όλα αυτά οδηγούν σε απαιτήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, απαιτήσει για την επιβολή φόρων, φόρο περιβάλλοντος, οικολογικό φόρο. Τώρα λοιπόν σούσει τη οικονομική κρίση στην Ευρώπη όλα αυτά τα βρίσκω τουλάχιστον ατυχή. Η διεύρυνση, της, η επέκταση τη οδηγία περί οικολογικού σχεδιασμού φοβάμαι ότι θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη γραφειοκρατία αντί ε, να ε, επιφέρει πλεονεκτήματα στους Ευρωπαίους πολίτες. Μία άλλη λεπτομέρεια που επιθυμώ να αναφέρω είναι η εξή. Αφορά σε εκείνο το σκέλος του εγγράφου όπου γίνεται λόγος για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης. Ε, βεβαίως ε, όλοι συμφωνούν ε, ως προς το ότι πρέπει να εγκαταλευτούν ε, οι ανοιχτές χωματερές ηχητά για τα απορρίμματα. Και εγώ το στηρίζω αυτό. Όμως αν λέμε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνεται κάψη σε ανοιχτούς χώρους ενταφιασμού ε, τότε ε, καταλαβαίνω ότι πρέπει να βρεθεί μια εναλλακτική λύση. Για όλους αυτούς τους λόγους δεν θα στηρίξουμε την έκθεση. Ε, θέλω να ζητήσω συγγνώμη που χτύπησα το σφυρί μου ε, που βιάστηκαν να το χτυπήσει ο συνάδελφος Ρώση για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αυτή η έκθεση είναι και πάλι ε, δήλωση προθέσεων που δύσκολα μπορούν να επιτευχθούν κυρίως επειδή ε, αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια κρίση οι συνθήκες και οι συμβάσεις που έχει υπογράψει το Συμβούλιο ή το Κοινοβούλιο είναι περιβαλλοντικής φύσεως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν μπορεί όμως να οδηγήσει στη φτώχεια ούτε τους πολίτες ούτε τις επιχειρήσεις, απλά και μόνο προς όφελος τρίτων χωρών. Έχουμε λοιπόν πολύ αυστηρές προδιαγραφές, οι τρίτες χώρε αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, ε, η μεταφορά λοιπόν αυτών των, ε, ε, η μεταγκατάσταση αυτών των επιχειρήσεων θα δημιουργήσει προβλήματα. Σε άλλες χώρες θα πάνε που δεν είναι τόσο αυστηρές οι Ευρωπαίοι πολίτες κάνουν και τη δουλειά τους και αυξάνονται και οι εκπομπές ε, στο περιβάλλον. Το να χάσει η Ευρώπη την ανταγωνιστικότητά της αυτό σημαίνει ότι θα διαρκέσει περισσότερο η κρίση. Γι' αυτό λοιπόν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος εμείς καταψηφίσαμε την έκθεση. Εάν τελικά με τις ε, σημαντικές τροπολογίες που θα κατατεθούν θα βελτιωθούν τα επίμαχα σημεία της έκθεσης έχοντας ε, κατά νου το, τη σφαιρικότερη έκθεση εμείς τελικά αντί για να καταψηφίσουμε, το πολύ πολύ να δηλώσουμε αποχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνάδελφε κύριε Ρώση. Ο συνάδελφος κύριος Χαρτούγκ για 1,5 λεπτό. Μιλάμε για την έκθεση μπράντι για την ε, αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων. Ο συνάδελφος μας ε, έχει παρουσιάσει ωραίες προτάσεις, αλλά ε, το κείμενο, ε, το, το νόημα είναι κενό. Δεν μας λέει τίποτε. Θέλ, μιλάει για την αποτελεσματικότητα των πόρων ανάλογα με τον κύκλο ζωής που αναφέρεται σε ένα πιο αισιόδοξο χρονοδιάγραμμα. Δεν ξέρω πού θέλει να καταλήξει με όλα αυτά ο κύριος Γκεμπράντη αυτό που θα συμβεί θα είναι να πάνε πολλά χρήματα, πολλά χρήματα στις τσέπες των φίλων του. Μας μιλάει για ένα φόρο, για τη χρήση χωματερών, για την πολιτική των αποβλήτων. Η Βαρόνη Άστον θα χρειαστεί να μεταβεί σύντομα στα κράτη-μέλη για να δει τι γίνεται με την ε, με τα απόβλητα και τα απορρίμματα αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να προστατεύσουμε τους φυσικούς πόρους, όλοι το γνωρίζουν αυτό. Δεν χρειαζόμαστε τις ε, ηλίθιες ε, υποδείξεις ε, του κυρίου Γκεμπράντη. Τι θα, το, τι θα την κάνουμε αυτή την έκθεση, διαρωτώ με. Αναφέρεται ο κύριο Γκεμπράντη σε κριτήρια για το τέλος της διάρκειας ζωής των αποβλήτων η έκθεσή του ανταποκρίνεται απόλυτα σε αυτό το κριτήριο. Θα πετάξω λοιπόν το, την έκθεσή του σε ένα καλάθι των αχρήστων. Συνάδελφε Χάρτουγκ, θα δεχτείτε μία ερώτηση από τον κύριο Γκεμπράνδη. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Χαρτόγκ δεν κατάλαβε πολύ καλά ποια είναι η κατεύθυνση που θέλω να ακολουθήσω. Είναι μια κυκλική κατεύθυνση. Ίσως δεν είναι απόλυτα σαφές και με κατηγορεί για τους στόχους που έχω αναφέρει για την προστασία του περιβάλλοντος. Όταν ο χαλκός για τον οποίο θέτω με 20 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ενώ ήταν το ποσό 6 δισεκατομμύρια πριν από 20 χρόνια, είναι αυτή αυτή, αυτό ένα πρόγραμμα για το περιβάλλον ή πρόκειται για κάτι το οικονομικό. Πώς το αντιλαμβάνεται ο ίδιος. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε για την απάντησή σας. Ήταν μάλλον όμως μια ερώτηση, αλλά ήταν μάλλον παρατήρηση. Είστε κλειστός, περαμένετε κλειστός σε ένα γυάλινο πύργο και κανείς δεν μπορεί να σας αγγίξει. Αυτό που ήθελα να πω στην παρέμβαση μου ήταν ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί με τους φυσικούς μας πόρους, αλλά όχι με τον τρόπο που προτείνετε εσείς. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, τώρα θα ακολουθήσουν οι επόμενοι ομιλητέ. Συνάλφο Ζήμπα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστώ τον εισηγητή, τον ε, κύριο Γκεμπράντη και το δικό μα τον σκιώδη εισηγητή, τον κύριο Φλόρεντ, που και οι δύο ε, κατάρτισαν μια πολύ καλή έκθεση. Επιτρέψτε μου μια ιστορική αναδρομή για να δούμε λιγάκι ε, ποιες, ποιοι είναι οι παράγοντε εκείνοι που οδήγησαν στην σημαντική πρόοδο τη Ευρώπη. Θέλουμε να παραμείνουμε σε αυτή την τροχιά. Ποια ήταν τα βασικά στοιχεία Νομίζω ότι ήταν αυτή η σημαντική αύξηση των πόρων. Ε, γύρω στο 1400 ε, περίπου είχε κανείς, ε, χρειαζόταν μισό εκτάριο στην Κίνα για την διατροφή μιας οικογένειας. Σήμερα όμως έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα εκτάρια. Ποιοι είναι οι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτό. Ο ανταγωνισμός που επικράτησε ανάμεσα σε διάφορα κράτη κατόπιν τούτου. Βλέπετε ότι υπήρξε αγώνας όλων όλων έναντι όλων. Υπάρχει γνώση στην Ευρώπη που την αποκτήσαμε και μπορούμε με λογική να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις και προσπαθούμε να ε, κυριαρχήσουμε στη φύση, ε, να γνωρίζουμε τους ε, φυσικούς νόμους και να τους χρησιμοποιούμε στην οικονομία. Τρίτον, υπάρχουν οικονομικές δομές, μάλλον δομές ιδιοκτησία στην Ευρώπη που προήγαγαν την ανάληψη ευθυνών με την έννοια ότι οι άνθρωποι πλέον νιώθουν ότι είναι υπεύθυνοι με αυτά που έχουν να συμβάλλουν στο γενικό γενικότερο καλό. Ε, κατόπιν κίνητρα, ε, τιμέ λοιπόν, τιμές ε, που να προκαλούν και να προσφέρουν κίνητρα. Όλη αυτή η πρόοδο βασίζεται στο σύστημα των τιμών και καταβάλλονται προσπάθειες να συμπεριλαμβάνεται και το εξωτερικό κόστος στου υπολογισμούς. Αυτό βέβαια είναι δύσκολο διότι σε τελική ανάλυση χρειαζόμαστε την πολιτική συνένεση εάν θέλουμε να επηρεάζουμε τεχνητά τις τιμές της αγοράς. Τρίτον, χρειαζόμαστε και ε, διατάξεις. Είναι σημαντικό να εκπονούνται διατάξεις μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην εφαρμογή και όχι ε, τόσο στο ε, να μεταθέτουμε το στόχο. Σε ευχαριστώ. τώρα. Ευχαριστώ. Η πολιτιστική πρόοδο επισπεύθηκε χάρη στην ευκαιρία απόκτηση ενέργεια. Ταυτόχρονα όμω είχαμε και εξάντληση ενεργειακών και άλλων πρώτων υλών. Αυξήθηκε αισθητά η κατανάλωση και η ευμάρεια των κοινωνιών. Η περαιτέρω αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού με το μέχρι τώρα καταναλωτικό μοντέλο δημιουργεί τεράστιε προκλήσει. Δεν μιλούμε μόνο για τα μέχρι τώρα προβλήματα και κλιματικέ ακλαγέ. Ε, αλλά για την ε, ορθολογική λύση και ε, αποτελεσματική αξιοποίηση των, ε, των πόρων μας με ένα άλλο καταναλωτικό μοντέλο προκειμένου να μπορέσουμε όλοι να απτυχθούμε ρωμανικά. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι έχουμε όλο και περισσότερη μεταποίηση πρώτων υλών με αυξημένη προστιθέμενη αξία. Γιατί πιστεύετε ότι η Κίνα θέλει να ε, μεταποίηση λαθανίδες ε, στη χώρα της. Ενώ το σύνθημα της Ρωσίας ε, πρώτες ύλε για εξυγχρονισμό είναι πλέον παροχημένο. Έχουμε μετακατάσταση ενεργειοβόρων ε, ε, βιομηχανιών εκτός της Ευρώπης, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να, να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους ορυκτούς ε, πόρους, δάση, εδάφη, νερά κτλ. Θα πρέπει να ε, κάνουμε οικονομίες, υλικές και τεχνολογικές αντικαταστάσεις, ε, ανακύκλωση, να αξιοποιήσουμε τους ε, ιδίους πόρους σε τοπικό επίπεδο Επίσης να δημιουργήσουμε οικονομικούς και φορολογικές προϋποθέσεις για να ανακτήσουμε την οικονομία μας στην Ευρωπαϊκή και την ανταγωνιστικότητά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να επισημάνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις, τις επιζήμιες δραστηριότητες πολυεθνικών εταιριών καθώς και τον οικονομικό προστατευτισμό ορισμένων χωρών που είναι και μέλη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου. Ευχαριστώ. Πολύ ωραίο, Άλφος Κράμερ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης τον συνάδελφο κύριο Γκέμπραντι για την πολύ καλή δουλειά που έκανε. Ε, πολλά από αυτά που αναφέρονται στην έκθεση εγώ τα στηρίζω. Είναι σωστό να λέμε ότι οφείλουμε να άρουμε τα εμπόδια στην κοινή αγορά, κυρίως όταν πρόκειται για την οικονομική διαχείριση των πόρων. Νομίζω λοιπόν πολλά από αυτά που ελέγχθησαν δυστυχώς ε, επίσης δεν είναι σωστά. Ε, χάρη δεν αυξάνεται η τιμή του χαλκού ε, γιατί μειώνονται τα αποθέματα χαλκού. Πολλές φορές δεν αυξάνονται οι τιμές ε, επειδή ε, φθήνουν οι πηγές, μόνο επειδή τυπώνεται πολύ χρήμα και επειδή δεν είναι πια σταθερά τα ομόλογα, αγοράζονται οι υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τις ε, πρώτες ύλε. Αυτή λοιπόν είναι η ανάλυση που πρέπει να γίνεται ότι όλα αυτά δεν έχουν ε, σχεδόν καμία σχέση με την, ε, τον περιορισμό των αποθεμάτων. Υπάρχουν ορισμένα θέματα στην έκθεση που τα βρίσκω λανθασμένα. Το ένα είναι έτοιμα επέκταση της οδηγίας περικολογικού σχεδιασμού. Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την αρχή ότι η καλύτερη λύση βρίσκεται μέσα από τον ανταγωνισμό. Εδώ στην περίπτωση αυτή αναφέρεται ήδη ε, το, το οικολογική υπαγόρευση. Επίσης ε, η Ευρώπη, στην Ευρώπη ε, δεν νομίζω ότι είναι σωστό να απαιτήσουμε νέους φόρους στη στιγμή που υπάρχει αυτή τη στιγμή η κρίση. Ευχαριστούμε κύριε Κράμερ. Θα δεχτείτε μία ερώτηση από την άλλη, κύριο Ζήμπα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, ο συνάδελφος Κράμαρ είπε ότι τυπώνουμε πολύ χρήμα, γι' αυτό αυξάνονται οι τιμές. Γνωρίζουμε ότι η Fed με τα quantitative easing programs ε, έχει τυπώσει χρήμα και ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν το πράττει αυτό. Μήπως έχετε εσείς πληροφορίες ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτή τη στιγμή τυπώνει υπερβολικές μεγάλες ποσότητες χρήματος. Κοιτάξτε, είναι θέμα πολιτικής αξιολόγησης. Να σας υπενθυμίσω, βέβαια όλα αυτά τώρα δεν έχουν καμία σχέση με το θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει απαντώ στην ερώτηση. Από Δεκέμβρη μέχρι Φεβρουάριο ένα δις ευρώ τυπώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ρευστότητα στις ε, χώρες του Νότου. Ε, το γεγονός ότι κινδυνεύει σταθερότητα, ε, αυτό νομίζω δεν ισχύει. Με την πολιτική αυτή απλά πιέζουμε την κατάσταση σχετικά με τις πρώτε ύλες. Σα είπα ότι ότι πολλοί επενδυτέ επενδύουν σε πρώτε ύλε ε, γιατί νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια και βεβαίω κερδοσκοπούν και με τι πρώτε ύλε. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Κυρία, κυρία Χάση, για δυόμιση λεπτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ Ευχαριστώ τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά του. Η βελτίωση της χρήσης αυτών των πόρων, παράγοντας μεγαλύτερη ευημερία με λιγότερους φυσικούς πόρους, είναι κάτι το αναπόφευκτο αν θέλουμε να εξελιχθούν ε, οι εξελιγμένες κοινωνίες μας να εξακολουθούν να ζούνε. Ο αρμόδιος ε, επίτροπος αντιμετωπίζει με σοβαρότητα αυτό το θέμα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Χαιρετίζουμε αυτή την πρωτοβουλία, αλλά είμαστε λιγότερο ικανοποιημένοι από το γεγονό ότι η Επιτροπή σε δύο χρόνια δεν μα έχει υποβάλει καμία συγκεκριμένη πρόταση για αυτό το θέμα. Παραδείγματο χάρη, η ανακύκλωση των ε, μεταλλικών συσκευασιών. Ε, υπάρχει ένα σύστημα υποδείξεων σε ορισμένες χώρες που θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί παντού. Ε, γιατί λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά στις χώρες όπου εφαρμόζεται, αλλά δεν έχει γίνει τίποτε. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος επιμένει πάρα πολύ στην ανάγκη ε, προσδιορισμού συγκεκριμένων στόχων που θα συνοδεύονται από δείκτες για να βλέπουμε κατά πόσον επιτυχάνονται ή όχι αυτοί οι στόχοι. Αυτό είναι αναγκαίο αν θέλουμε κάτι να συμβεί. Αν θέλουμε δηλαδή όλα αυτά να μην παραμείνουν απλώς λόγια και να είναι επίση πολύ σημαντικό να περιορίσουμε την, την κατανάλωσή μας πρώτων υλών με απόλυτο τρόπο. Δεν αρκεί να, να γίνεται χρησιμοποίησή τους κατά τη διάρκεια της παραγωγής αν έχετε αύξηση σε απόλυτους αριθμούς της κατανάλωσης. Χρειαζόμαστε λοιπόν πάρα πολλά πράγματα κυρίως να βελτιώσουμε τη διαδικασία της ανακύκλωσης. Είναι αντιφατικό και τελείως τρελό το ότι έχουμε θαυμάσεις πολιτικές δηλώσεις με έκφραση ανησυχίας για τη διαθεσιμότητα εδαφών και τι γίνεται με την ανακύκλωση. 1% είναι το ποσοστό. Λιγότερο από 1% οι ηλεκτρικές συσκευές. Σε αυτές βρίσκουμε 15% παραπάνω ε, υλικά από ό,τι σε κάποια ορυχεία. Τα κινητά τηλέφωνα ε, μπορούν να, από, τα, από τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να πάρουμε ε, ένα πολύ σημαντικό αριθμό 15 τόνους, 15 τόνους από διάφορα πολύτιμα υλικά στη Φιλανδία αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα, τις συνέπειες, ε, τις περιβαλλοντικές, τις εκπομπές, οι οποίες είναι δέκα φορές υψηλότερες από αυτά που είχαν προβλέψει οι άδειε. Είναι λοιπόν απαραίτητο να βελτιώσουμε τη διαδικασία της ανακύκλωσης, ώστε να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις αυτής της διαδικασίας. Ευχαριστούμε κύριε Χάση. Κύριε Ρόσμπαχ τώρα. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, έχουμε εγκρίνει πολλές ε, εκθέσεις που στόχο έχουν την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων, ε, περιορίζοντας ε, η δυνατότητα κατανάλωση. Αναλάβαμε την πρωτοβουλία για ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία για μια αιφόρο αξιοποίηση των κοινών μας πόρων. Γιατί όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποφασίζει πώς ε, τα κράτη-μέρη θα αξιοποιήσουν πιο αποτελεσματικά τους δικούς τους ενεργειακούς πόρους. Στην έκθεση περιλαμβάνονται πολλές προϋποθέσεις ό,τι αφορά την διαχείριση των αποβλήτων. Κατά τη γνώμη μου, το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων είναι εθνική υπόθεση. Δεν θα πρέπει να υπαγορεύεται από μια κοινοτική έκθεση. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εθνικές, τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες και συνθήκες. Επίσης μιλήσαμε για την σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων. Πολύ καλή πρόταση αυτή, αλλά υπάρχουν και άλλα κριτήρια. Δεν θα μπορέσω να υπερψηφίσω την έκθεση, παρόλο που έχει κάποια θετικά στοιχεία όπως πρόσβαση στα επιστημονικά πορίσματα για να γίνει μια ορθολογική αξιοποίηση των πόρων τελικά ίσως αντί να καταψηφίσω κρατήσω απλώς τα αποχής ε, λόγω και των θετικών σημείων. Θέλουμε να γίνει όλο και πιο φιλοπεριβαλλοντική νομοθεσία. Δεν αναφέρθηκε και η εξαγωγή απορριμμάτων, κυρίως πλαστικών απορριμμάτων προς τρίτες χώρες. Θα πρέπει κάτι τέτοιο να γίνει μια τέτοια ρύθμιση να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αποφύγουμε με την κατάσταση επιχειρήσεων. Ευχαριστούμε κυρία Ρόσπαχ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε την κυρία Ρόσπαχ. Ακολουθεί ο η ε, μπράσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, για να αντιμετωπίσουμε επίγοντα προβλήματα, ανεργία, την πληθωρισμό και την έλλειψη δημόσιων πόρων πρέπει να βρούμε νέους τρόπους να χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά τους πόρους που διαθέτουμε. Βεβαίως πρέπει να χρησιμοποιούμε τα δευτερογενή ε, ε, υλικά ε, με αποτελεσματικό τρόπο για να περιορίσουμε τα απόβλητα. Η βιώσιμη κατανάλωση πρέπει να αποτελέσει μια προτεραιότητα των ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων η μείωση των αποβλήτων, καλύτερη συγκέντρωση και επιλογή των αποβλήτων είναι ο μόνος τρόπος για την προστασία του πλανήτη μας. Καλύτερη, πιο βιώσιμη χρήση όλων των πόρων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πράσινη οικονομία. Η Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες που διαθέτει για να οδηγήσει όλα τα κράτη προς τη σωστή κατεύθυνση και να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για τις μελλοντικές γενιές πρέπει να αξιοποιούμε τους πόρους μας έχοντας εις υπόψη τις δυνατότητες της πραγματικές του πλανήτη μας. Επόμενος ομιλητής, Βέρτμαν, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ε, κρίση που διαρκεί καταδεικνύει ότι στην Ευρώπη πρέπει να αναζητήσουμε νέες δυνατότητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ανοιχτή οικονομία επεκτείνεται και η ζήτηση για θέσεις εργασίας μπορούν, μπορεί να καλυφθεί από τον τομέα της, των παραγωγικών πηγών. Οφείλουμε λοιπόν να ασχοληθούμε περισσότερο με τομεί που δεν τους έχουμε λάβει υπόψη μας, ε, όπως με τη δημογραφική εξέλιξη και την αυξανόμενη ζήτηση για τρόφιμα. Εγώ λοιπόν ε, κατόπιν τούτου συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει ε, ε, μια σωστή μεταχείριση της συζήτηση για τρόφιμα και των πρώτων υλών. Επίσης πρέπει να ασκηθούν έλεγχοι, να υπάρχει διαφάνεια αλλά και να προσφέρονται και εξηγήσει στους πολίτες μας. Αυτά πρέπει να αναφέρονται. Οι δικοί μας οι πολίτες είναι πρόθυμοι να συμβάλλουν ενεργά και το ίδιο ισχύει και για τους εθνικούς πολιτικού σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ του συναδέλφου για την έκθεσή του. Ευχαριστούμε, συνάδελφε Μπέρτμαν. Ο συνάδελφο Φράνκο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον συνάδελφο για την ποιότητα της έκθεσή σου που θα την υποστηρίξω με μεγάλη χαρά. Αγαπητοί συνάδελφοι, η οικονομία και η βιομηχανία μας στην Ευρώπη εξαρτώνται από πόρους και πρώτες ύλες που, σε χώρες που είναι όλο και περισσότερο ασταθείς και ο εφοδιασμός μας ε, ε, δεν είναι εξασφαλισμένος ας πούμε, τις, αν πάρουμε τις φανεριές που είναι απαραίτητε για τις ε, νέες τεχνολογίες και που τις ελέγχει απόλυτα η Κίνα. Για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας στη βιομηχανική και το προστατεύσουμε το περιβάλλον μας πρέπει να μάθουμε να εξαρτώμαστε λιγότερο από αυτούς τους πόρους αναπτύσσοντας καινοτόμους ε, ε, λύσεις και ανακύκλωση. Πρέπει να προχωρήσουμε προς μια κυκλική οικονομία στην οποία η παράταση της διάρκειας ζωής των υλών θα αποτελέσει προτεραιότητα από το στάδιο της σύλληψης και της δημιουργίας των προϊόντων μέχρι της επανάχρησης και της ανακύκλωσης των αποβλήτων και απορριμμάτων. Η ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων πρέπει επίσης να ενισχυθεί. Επίσης πρέπει να στραφούμε προς την βιώσιμη ε, εκμετάλλευση πόρων των οποίων η σημασία υποτιμάται. Είναι πρέπει να λάβουμε υπόψη το κεφάλαιο που αποτελούν τα δάση μιλάμε για μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και ένα θαυμάσιο ε, οικοδομικό υλικό. Απέναντι στο δυναμισμό των αναδιωμένων οικονομιών πρέπει να, είμαστε, να επιδείξουμε μεγαλύτερη φαντασία στη χρήση των πόρων ώστε να βρούμε την οδό, ξαναβρούμε την οδό της ανάπτυξης. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παροτρύνει τις επιχειρήσεις να δημιουργούν ε, προϊόντα πιο καινοτόμα και πιο βιώσιμα Υποστηρίζω τα πειράματα που γίνονται για την ε, περιβαλλοντική παρουσίαση των προϊόντων ώστε να ενημερωθούν σωστά και με αξιόπιστο τρόπο για τις, για περιβαλλοντικές επιλογές τους όταν αγοράζουν καταναλωτικά είδη. Το νερό είναι πολύτιμο αγαθό, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ευχαριστούμε συνάδελφε κύριε Φράγκο. Ο κύριος Κούτας για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, τα 12 τελευταία χρόνια βιώσαμε μια σημαντική αύξηση της τιμής των πρώτων υλών σε διεθνές επίπεδο, αλλά και μια ε, τάση προς την κερδοσκοπία. Και αυτό με τίμημα την, ε, τα προβλήματα που αντιμετώπισαν ε, εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών μας λόγω της κακής κατανομής των πόρων και της κερδοσκοπίας των αγορών. Γι' αυτό πρέπει να προωθήσουμε ένα ε, παγκόσμιο σύστημα για τους ε, φυσικούς σπόρους και καλό την Επιτροπή να συμπεριλάβει τους περιβαλλοντικούς κανόνες και τους κανόνες της, ε, του δίκαιου εμπορίου στην ημερήσια διάταξη του ΠΟΗ. Οι προσπάθειές μας πρέπει να συνεχιστούν για να ε, καταργήσουμε τους δασμούς για την εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών για να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους σπόρους μας. Τέλος, θα ήθελα να θυμίσω ότι η κερδοσκοπία ε, στις πρώτες ύλε έχει αρνητικές επιπτώσεις για τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών μας και γι' αυτό πρέπει να απογορεύσουμε, αυτή την πρακτική απλά και μόνο. Σας ευχαριστώ κύριε Κούτας, ο κύριος, η κυρία Μάνερ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, Επίτροπε, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτή την εξαιρετική έκθεση. Νομίζω πως όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε με τα όσα λέτε και χαίρομαι διότι μέσα σε αυτή την έκθεση παρατηρούμε και επιμένουμε για την ε, νέα χρήση των ανακυκλωμένων προϊόντων, των ανακυκλωμένων υλικών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό γιατί ξέρουμε πως στην Ευρώπη υπάρχουν χώρες όπου 100% όλα πάνε ε, στην ε, ε, στα απορρίμματα και δεν ανακυκλώνεται τίποτα. Είναι πάρα πολύ καλή λοιπόν η έκθεση αυτή. Πρέπει να επιμείνουμε για τα απορρίμματα, τα τροφικά απορρίμματα. Σε αυτή την έκθεση Γκερμπράντι επίσης υπογραμμίζεται η βιώσιμη χρήση των πόρων, ιδιαίτερα των δασικών πόρων. Είναι σημαντικό να επιμείνουμε για την καλή χρήση των ε, δασικών πόρων, γιατί το ξύλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την κατασκευή διαφόρων προϊόντων. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μάνερ. Για δύο λεπτά ο κύριος Μποτικόφερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Επίτροπε, κύριε Συγητά, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω ρητά τον κύριο Γκέρμπραντι για την έκθεσή του το μήνυμα που θα πρέπει να βγει από τη σημερινή συζήτηση για την κοινή γνώμη, για την οικονομία και για τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι ότι υπάρχει ισχυρή συνεργασία Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίως του κυρίου Ποτότσνικ και του Κοινοβουλίου σε θέματα εξοικονόμησης και αποτελεσματικής χρήσης των πόρων. Νομίζω ότι εδώ και πολύ καιρό γνωρίζουμε όλοι τα αποφασιστικά δεδομένα. Γνωρίζουμε η Ευρώπη ότι εξαρτάται όλο και περισσότερο από την ε, εισαγωγή ε, πρώτων υλών, περισσότερο από άλλες ύλες. Επίσης, θα ήταν μεγάλη βοήθεια για τη δυναμική της οικονομίας να προχωρήσουμε, να προωθήσουμε αυτή την εξοικονόμηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα έχει προϋπολογίσει. Μέχρι 3 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε εάν πάρουμε σοβαρά αυτό το θέμα υπόψη. Όλα αυτά που τα ξέρουμε, τι τα κάνουμε. Ε, εδώ θα πρέπει να δράσουμε. Η διακυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, αλλά κυρίω τα κράτη-μέλη και η ιδιωτική οικονομία και άλλοι φορεί θα πρέπει να συνεργαστούν με τρόπο λογικό. Και εκεί χωλαίνει η υπόθεση. Α είμαστε ειλικρινεί. Δεν ξέρω εάν ο κατάλογος μου δεν είναι πλήρης, αλλά μέχρι τώρα βρήκα τέσσερα κράτη-μέλη όπου Υπάρχουν κάποια σχέδια. Ε, ε, η Ολλανδία από το 10, η Αυστρία από τον Ιανουάριο ε, και η Μεγάλη Βρετανία και η Γερμανία αυτό το χρόνο. Η Γερμανία έχει φτάσει να το συζητάει και σε επίπεδο υπουργών. Καλά. Και στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος δεν εδέησαν να συζητήσουν τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρά τις μπλόκαραν. Ας είμαστε λοιπόν και φιλόδοξοι και σαφείς για να στείλουμε το μήνυμα. Τολμήστε να αναλάβετε την ηγετική θέση ή δώστε ένα παράδειγμα ή εν περιπτώσει αδειάστε μας στη γωνιά αν δεν μπορείτε. Ευχαριστώ. Τώρα για ένα λεπτό η κυρία Γιανακουδάκη. Thank you. Currently the... Σας ευχαριστώ. Αυτή τη στιγμή ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης ε, παράγει γύρω στους 6 τόνους ε, ε, απορριμμάτων. Αυτό είναι απαράδεκτο και γι' αυτό και υποστηρίζω κάθε μέτρο ανακύκλωσης και εκ νέου χρήσης. Έχουμε προχωρήσει πολύ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο το 40% των οικιακών αποβλήτων ανακυκλώνεται σε σχέση με το 11% πριν από 10 χρόνια. Έχουν γίνει πολλές προτάσεις στην πρόταση Μπράντι, αλλά συμπεριλαμβάνονται και κάποιες μη πρακτικές συστάσεις όπως η γενική απαγόρευση των ε, ε, υπαίθριων ε, των χωματερών. αυτό το σώμα πρέπει να γνωρίζει πως η φορολογία δεν είναι η λύση για κάθε πρόβλημα γιατί προτείνεται και η φορολόγηση των υπερβολικών απορριμμάτων. πρέπει να θεσπίσουμε ρεαλιστικούς στόχους με σταδιακή ε, αλλαγή από τις ε, χωματερές και αυτές οι αποφάσεις να λαμβάνονται σε επίπεδο κρατών μελών. Ευχαριστώ κύριε Γιανακουδάκη. Τώρα ο κύριος Σιμάνσκι. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την προσοχή σας ότι εδώ μιλάμε για μείωση κατά 95% των αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με το 1990. Αυτό είναι εξαιρετικός στόχος. Αλλά η μείωση της ε, ενέργειας που καταναλώνουμε είναι δύσκολο εγχείρημα. Η Πολωνία, η χώρα μου έκανε πολλά για να μειώσει το διοξίδιο του άνθρακα στις εκπομπές. Και οι προσπάθειες των κρατών μελών θα πρέπει να αναγνωρίζονται. Πρόκειται για την ε, ανάπτυξη στην Ευρώπη, άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τους στόχους και τις συνεχείς μειώσεις. Ούτε μας επιτρέπεται να είμαστε απλοϊκοί. Είπα, η Κίνα η Ινδία ε, έχουν τη μεγαλύτερη, το περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα και δεν μας ακολουθούν. Ευχαριστώ. Κυρία Γκαρντίν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλάμε για το συνδυασμό της προστασίας του περιβάλλοντος με την οικονομική ανάπτυξη που σίγουρα είναι ένα κεντρικό ζήτημα και αντιμετωπίζει μεγάλη, βρίσκει μάλλον μεγάλη συνένεση σε διάφορα επίπεδα. Η καλύτερη χρήση των πόρων παίζει τον πρώτο ρόλο και σίγουρα είναι δικό μας καθήκον να εγγυηθούμε μια ανάπτυξη που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σημερινών γενεών αλλά χωρίς να ε, εμποδίζει τις επόμενες γενναίε από το να ικανοποιήσουν τις δικέ τους ανάγκες. Ωστόσο, νομίζω πως πρέπει να προωθήσουμε εδώ μια ολόκληρη νοοτροπία. Ε, γι' αυτό και πιστεύω πως θα πρέπει να αποφύγουμε αυτόν τον ε, κάπω καθοδηγητικό τρόπο και τόνο της έκθεσης αυτής που τονίζεται και από τον εισηγητή. Πολλά πράγματα ήδη υπόθηκαν. Με ανησυχία, για παράδειγμα, η μεταφορά από την εργασία στην απασχόληση. Η έλλειψη ενός μιας αξιολόγησης αντικτύπου και σε οικονομικό επίπεδο μπορεί να έχει ως μοναδικό αποτέλεσμα την επιδίνωση την ήδη, το, του ήδη μεγάλου φορολογικού φόρτου ε, στους, ε, για τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν νομίζω πως είναι δικό μου καθήκον αν θα πρέπει να τρώνε ναι ή όχι ε, ζωικές πρωτεΐνες. Νομίζω πως είναι μάλλον ε, πιο ενδιαφέρον τα όσα έχει ήδη πει το Ευρωκοινοβούλιο εκφράζοντας ε, τη γνώμη του κατά της ε, σπατάλης των τροφίμων. Ελπίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε πιο επικοδομητική προσέγγιση και ρεαλιστική. Θα πρέπει να στηρίξουμε κυρίως τις προτάσεις που στόχο έχουν να διευκολύνουν την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις καινοτόμες τεχνολογίες, να στοχεύσουμε στην έρευνα και στην καινοτομία, αλλά να δουλέψουμε και με την βοήθεια του παραγωγικού κλάδου που μας δίνει αξιόπιστα στοιχεία για τις πόρους που βασίζονται όχι μόνο σε οικονομικές αξιολογήσεις, αλλά και σε επιστημονικές γνώσεις. Και έπειτα χρονική στιγμή. Όποιος βιάζεται σκοντάφτη λέμε στην Ιταλία και γι' αυτό προσοχή να μην βιαστούμε πολύ. Κυρία Γκαρδίνη μου, επιτρέπετε ερώτηση του κυρίου Μπουτικόφερ. Επιτικόφερ. Κύριος Μπουτικόφερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία συνάδελφε, για να καταλάβω τι εννοείτε αν το προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή φορολόγηση της εργασίας να μειωθεί και να αντικατασταθεί από φορολόγηση των φυσικών πόρων. Ε, πώς αυξάνεται η επιβάρηση των πολιτών, γιατί εγώ δεν το κατάλαβα. Και μια δεύτερη ερώτηση. Αν είναι γεγονός και ισχύει ότι η παραγωγικότητα στην εργασία αυξήθηκε σημαντικά από την παραγωγικότητα των πόρων, γιατί εμποδίζουμε τη βιομηχανία αντί να προωθήσουμε και την παραγωγικότητα των πόρων. Η κυρία Γκαρντίνη. Εγώ πιστεύω πως όταν ε, μιλάμε για φόρους δεν είδαμε ακόμα φόροι, ένας φόρος να καταργεί κάποιον άλλον και έπειτα πιστεύω πως ε, η φορολογία και είμαι υπέρ της επικουρικότητας μέχρι στιγμής είναι αρμοδιότητα της ε, εθνική και δεν πιστεύω πως Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε εκ των άνω τέτοιου είδους ε, φορολογήσεις. Ε, περισσότερο θέλουμε να αλλάξουμε την οτροπία των ε, πολιτών. Το να θέλουμε να επιταχύνουμε υπερβολικά κάποιες ε, διαδικασίες και θετικές με στάδια πολύ στενά μεταξύ τους, αυτό έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά ο κύριος Γκρότη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Συγητά, σκιώδης εισηγητές. Το πνεύμα πρόθυμο, αλλά η σάρξ ασθενής. Ταιριάζει αυτό στην ορθολογική χρήση των πόρων. Όλοι θέλουν το σωστό, αλλά πώς να το κάνουν. Εθελοντικά μέτρα είχαμε και στην αυτοκινητοβιομηχανία και αλλού και απέτυχαν παταγωδός. Τώρα η αποτελεσματική χρήση των πόρων η φιδό στη χρήση των πόρων αφορά την υγεία, την παιδεία, την οικονομία, τη γεωργία. Ε, ισχύει για όλους τους τομείς της οικονομίας μας. Αν ε, δούμε, ας πούμε, ε, το συμβούλιο, προς την κατεύθυνση του Συμβουλίου, βλέπω ότι απέχει, αλλά εκείνο είναι χαμένο, γιατί είναι πολύ καλή η έκθεση Μπράντι. Το θέμα θα μας απασχολήσει εδώ, ε, για καιρό ακόμη και θα κρίνει αν θα ζήσουμε στο μέλλον σε ευημερία στην Ευρώπη και τι περιβάλλον θα έχουμε στην Ευρώπη. Και βεβαίως ε, εδώ σημαντική είναι, σημαντικά είναι τα μέσα. Εξωτερικοποίηση του εσωτερικού κόστου. Αυτό θα πρέπει να γίνει, δεν γίνεται αλλιώ. Δηλαδή όποιος ε, ρηπαίνει αέρα, νερά πρέπει να πληρώνει. Σήμερα γίνεται μέσα από τις, ασφαλισ... τις ασφάλειες υγείας. Ε, θα πρέπει όμως να ε, πληρώνουμε με τους φόρους μας. Χρειάζεται λοιπόν εσωτερικοποίηση και γι' αυτό απαιτείται θάρρος. Μόνο έτσι θα ανταποκριθούμε στις μελλοντικέ και τις τωρινές δηλαδή προκλήσεις. Αύξηση του πληθυσμού του κόσμου στην Ευρώπη, μείωση, τεράστιες προκλήσεις και γι' αυτό η έκθεση Γκερμπράντι είναι πολύ καλή εκκίνηση για να σκεφτούμε νέες πολιτικές. Και Κομισιόν θα πρέπει να σκεφτόμαστε ε, μακροπρόθεσμα, να δούμε όλο τον κύκλο της ζωής, να δούμε και το εργοστάσιο που κατασκευάζεται το αυτοκίνητο. Εκεί σέβονται τους πόρους, τους χρησιμοποιούν σωστά. Παντού πρέπει να επιδείξουμε θάρρος στα μέτρα που θα λάβουμε και να μην επιμένουμε στο status quo, γιατί θα το πληρώσουμε ακριβά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκρότε. Τώρα η κυρία Τσανόνη. Συγχαίρω τον κύριο Γερμπράντη για την εξαίρετη έκθεση. Η μετάβαση προ μια αποτελεσματική οικονομία στην χρήση των πόρων είναι αναπόφευκτη και απαραίτητη. Το 2050 ο παγκόσμιο πληθυσμό θα φτάσει τα 9 δισεκατομμύρια ανθρώπου και καθένα από αυτού θα θέλει καλύτερη ζωή. Όπω υποδεικνύει η Κομισιόν, στο σημερινό ποσοστό εκμετάλλευση των πόρων, ε, το 2050 θα χρειαζόμαστε δύο πλανήτε αντί γη για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον παγκόσμιο πληθυσμό τον προσαρμόσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική σε καλύτερη χρήση λοιπόν των πόρων είναι απαραίτητη οικονομική προϋπόθεση. Θα πρέπει να αρθεί κάθε φραγμός στην αγορά ανακύκλωσης και νέας χρήσης των αποβλήτων και πρέπει να προωθηθούν οι, διαδικασίες για τη συλλογή, συγκομιδή και νέα χρήση των αποβλήτων. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε για δείκτες για τη χρήση των πόρων, την οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή δηλαδή το αποτύπωμα στη γη, το, αποτύπωμα το ιδωτικό και στον άνθρακα επίσης. Αυτοί οι δείκτες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να προωθηθούν νομοθετικές πρωτοβουλίες για την βιώσιμη ανάπτυξη και για την καλύτερη χρήση των πόρων. Ευχαριστώ κύριε Τζανόνι και τώρα ο κύριος Σιμάνσκι. Για ένα λεπτό. Μια ισορροπημένη πολιτική πρώτων υλών θα πρέπει να εδράζεται σε τρεις πυλώνες. Αποτελεσματικότητα, ανακύκλωση και καλή αξιοποίηση των πόρων. Δυστυχώς αυτή η ισορροπία δεν υπάρχει στην έκθεση που έχει υποβληθεί. Πρόκειται για την αποτελεσματικότητα κυρίως. Όταν όμως μιλάμε για την πολιτική των ε, πρώτων υλών θα πρέπει να δούμε και άλλα μέτρα και άλλους φόρους, όχι μόνο των πρώτων υλών. Η υπεραξία ε, που θα φορολογείται θα επηρεάσει όλο το σύστημα. Αυτό βέβαια επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της ε, ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Μία πρόσθετη φορολόγηση των πρώτων υλών τη θεωρούμε απαράδεκτη. Πρέπει κυρίως να μας απασχολήσει το μέλλον, η ανάπτυξη στο μέλλον. Νομίζω ότι η έκθεση δεν ανταποκρίνεται στις μεγάλες προσδοκίες της ομάδας μου και γι' αυτό δεν μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σιμάνσκι και τώρα για δύο λεπτά η κυρία Ήμπνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά, όμως θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα βασικά σημεία. Υπέβαλα και τροπολογίες, διότι πιστεύω ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους μας. Ό,τι κάνουμε πρέπει να προσανατολίζεται στην οικονομική ανάπτυξη. Είναι αυτονόητο ότι Πολύ σημαντική είναι και η πράσινη οικονομία, αλλά σε εποχές κρίσης δεν μπορούμε να αυξάνουμε τις διοικητικές δαπάνες. Ας πούμε, απαγόρευση των χιτά. Αν προχωρήσουμε στην απαγόρευση θα πρέπει να δούμε πρώτα μήπως μπορούμε να αξιοποιήσουμε όντως διαφορετικά τους σπόρους. Δεν νομίζω ότι ενδείκνυνται οι εποχές για επιβολή νέων φόρων. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε. Τώρα, για το ζωικό λεύκομα είναι δύσκολο να προσανατολίσω με την παραγωγή. πιστεύω επίσης ότι οι πραγματικές τεχνικές δυνατότητες θα πρέπει να μας προσανατολίζουν πάντοτε. Από εκεί ξεκινάμε. Ούτε μπορούμε να μειώσουμε την ποσότητα των αποβλήτων, πιστεύω, όπως αναφέρει, τόσο όσο αναφέρει και προβλέπει ο εισηγητής. Επίσης, οι πληροφορίες και η ενημέρωση του τελικού καταναλωτή είναι πολύ θετικό πράγμα. Πρέπει όμως να είναι ε, έξυπνες κατανοητές. Υπάρχουν στην έκθεση ορισμένες σημαντικές ε, παρατηρήσεις ε, και προτεραιότητες. Λείπει όμως η αναφορά στην κρίση που μαστίζει τώρα την Ευρώπη. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να δούμε πώς θα δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας επίσης για τη δική μας τη γενιά και για τις επόμενες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Χίμπνερ. Ενάμιση λεπτό. Ε... Η κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αποτελεσματική χρήση και η εξοικονόμηση πόρων πρέπει να αυξηθεί για να μπορέσουμε να επιτυχάνουμε περισσότερα με λιγότερες πρώτες ύλες. Έτσι θα δημιουργηθούν και θέσεις απασχόλησης και θα έρθει και ανάπτυξη μακροπρόθεσμα. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ ε, σημαντικό το θέμα αυτό για την ανταγωνιστικότητα. Η έκθεση ποντάρει κυρίως στην καινοτομία και την έρευνα. Επίσης, ε, έρχεται να διαπιστώσει ότι οι κρατικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις ε, σε ρηπαίνουσες δραστηριότητε πρέπει να τερματιστούν. Καλό είναι αυτό. Θα πρέπει να επενδύσουμε αλλού, στην έρευνα και στη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Θέλουμε ε, να έχουμε μια σαφή στρατηγική. Η ε, αποτελεσματική χρήση των πόρων συνδέεται άμεσα με τον ανεφοδιασμό σε πρώτε ύλε. Εξαρτόμαστε και για τα ορυκτά και για τα μαέταλα και για γενικότερα πρώτες ύλες και είμαστε εισαγωγής θα πρέπει να προχωρήσουμε και να προωθήσουμε την έννοια του urban mining, δηλαδή να χρησιμοποιούμε πρώτες ύλε που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα τις ε, ανακυκλώνουμε, θα τις χρησιμοποιούμε με τρόπο ευφύ. Γι' αυτό θεωρώ την έκθεση πάρα πολύ καλή για τη συνέχιση ε, των ε, συζητήσεων προς την κατεύθυνση αυτή. Από την άλλη όμως είναι πολύ σαφές ότι η μετατόπιση της φορολογίας από την εργασία ε, στο περιβάλλον χρειάζεται περαιτέρω σύντηση. Ευχαριστώ για ένα λεπτό η κυρία Γκέρλινγκ. Thank you, President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πέρσι η ομάδα μου καλωσόρισε, τόσο τον οδικό χάρτη του Κομισιόν όσο και τα απορίσματα του Συμβουλίου για την ε, ε, αποτελεσματική χρήση των πόρων το Δεκέμβριο. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι είναι θετικές οι εκθέσεις αυτές ε, της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω λοιπόν τον εισηγητή, ωστόσο νομίζω ότι πρόκειται για έναν ε, κατάλογο, ένα μάλλον ευχολόγιο, το οποίο είναι και λίγο ασυνάρτητο. Υπάρχουν πολλοί τομείς που δεν μπορώ να συμφωνήσω μεταξύ αυτών ο περιβαλλοντικός φόρο. Ε, ε, υπονόησε ότι η γεωργία είναι μόνο, έχει μόνο αρνητικό αντίκτυπο και η έλλειψη ορισμού ε, για πάρα πολλά θέματα όπως το βλαβερό περιβάλλον ή οι επιδοτήσεις. Λυπούμε λοιπόν που αυτή η μπήκε σε χωράφια τα οποία βρίσκουν αναπαράδεκτα η, δικιά, η δική μας Βρετανική Συντηρητική Παράταξη. Σας ευχαριστώ κυρία Γκέρλινγκ. Η κυρία Κόρχολα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως λέει και η πρόταση ψηφίσματος, αντιμετωπίζουμε μεγάλες προκλήσεις για το περιβάλλον. Γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να δρούμε μακροπρόθεσμα. Είναι πολύ σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώς τόνισε την αποτελεσματική χρήση των πόρων και στη στρατηγική της Ευρώπη 2020. Η αύξηση του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο οι ανάγκες ε, για παραγωγή τροφίμων σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό μας οδηγεί σε μια κατάσταση ε, που θα πρέπει από σήμερα να προετοιμαστούμε για τη βιώσιμη ανάπτυξη του μέλλοντος. Η σημερινή απάντηση και η σημερινή απόφαση είναι πολύ κρίσιμη. Θα πρέπει να αξιοποιούμε καλύτερα τους πόρους, να τους εξοικονομούμε για να έχουμε μια οικονομία πολύ πιο αποτελεσματική. Αυτό θα ενισχύσει και τη βιομηχανία μας παγκοσμίω. Ωστόσο θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν σχεδιάζουμε τα μέτρα που λαμβάνουμε. Έτσι ώστε να χρησιμοποιούμε τους πόρους όσο γίνεται με πιο αηφόρο και βιώσιμο τρόπο. Για το λόγο αυτό δεν είμαι βέβαια ότι χρειαζόμαστε νέες νομοθετικές προτάσεις. Πιστεύω ότι το αντίθετο χρειάζεται να προσέξουμε γιατί θα πρέπει να ε, υλοποιείται καλύτερα και να εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία και είναι και περίπλοκη η νομοθεσία με επικαλύψεις και ο Πρόεδρος. Δεν ήθελα να σας διακόψω, αλλά θα πρέπει να μιλάτε πιο αργά, γιατί δεν σας προλαβαίνουν οι διερμηνείς. Και μου στέλνουν μηνύματα εδώ ότι δεν μπορούν να σας παρακολουθήσουν. Ε, επιπλέον, η πρόταση ψηφίσματος ε, είναι υπερβολική. Ε, γιατί είναι πραγματικά ε, ενιαία αντιμετώπιση για όλους, αλλά η κατάσταση δεν είναι ενιαία. Ε, διαφέρει από χώρα σε χώρα. Στο βορρά η αποτέφρωση ήταν και ε, αποτελεσματική και αναγκαία γιατί ε, δημιούργησε ενέργεια. Και η φορολογία δεν βοηθάει ενιαία όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα τη Βόρεια Ευρώπη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φλόρενς και ως σκιώδη συγκητή για την ομάδα μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Κόρχορα. Ορίστε, σας έμεινε και χρόνος. Αν θέλετε όλοι οι Ευρωπαίοι να καταλαβαίνουν αυτά που λέτε, σας παρακαλώ μην τα διαβάζετε με ταχύτητα φωτός. Και επίσης να έχουμε τη δυνατότητα, αν διαβάζετε κείμενα έτσι κι αλλιώς, να τα δίνετε προηγουμένως στους διερμηνείς για να τους διευκολύνετε. Ο κύριος Λάινεν, για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, συνηθίζεται να διαβάζονται για 1,5-2 λεπτά τα κείμενα. Είναι άσχημο αυτό, έπρεπε να μιλάμε ελεύθερα. Κύριε Ποτότσνικ, εσείς ε, τον τη χάρτη πορείας για το 2050 το παρουσιάζετε σωστά ως μετασχηματισμό παραγωγής, κατανάλωσης, οικονομίας. Και για το μεγάλο μετασχηματισμό χρειάζονται όλοι οι δρόντες, όλα τα επίπεδα. Καλό είναι που στις Βρυξέλλες υπάρχει μια πλατφόρμα αποτελεσματικής χρήσης των πόρων και παρόμοιο πρέπει να γίνει και στα κράτη-μέλη, στις περιφέρειες, μέχρι κάτω στις, στους Δήμους και τις κοινότητες. Ε, υπάρχει σχετικό πρόγραμμα. Ο κ. Μπουτικόφερ ε, ρώτησε για προγράμματα αποτελεσματικότητας των πόρων. Το ίδιο θέμα. Έχουμε τα ΝΑΠΑ στα ΝΑΜΑΣ, ε, προγράμματα προσαρμογής, μετριασμού στην αλλαγή του κλίματο. και εδώ θα πρέπει να κάνουμε παρόμοια προγράμματα για την αποτελεσματική χρήση των πόρων που θα τα πάρουν τα κράτη-μέλη. Επίσης ε, υπάρχουν και όλα τα άλλα χαρτοφυλάκια ε, ε, οικονομικών, οικονομικά συμπερίληψη εξωτερικού κόστου στο φορολογικό μας σύστημα. Πώς θα κερδίσουμε με το μέρος μας τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών γιατί χρειάζεται καινούριο μοντέλο το οποίο θα επενεί και θα επιβραβεύει την αηφορία και τη βιωσιμότητα και όχι την υπερβολική κατανάλωση. Ευχαριστώ κύριε Λάινεν. Α, συγγνώμη. Μπλε κάρτα από την κυρία Μέρκη. Ενδιάμεση ερώτηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συνάδελφε Λάιν, μιλήσατε για νέα επιχειρησιακά μοντέλα, αλλά ε, το θέμα δεν είναι πάντα η τεχνολογία και τα νέα μοντέλα των επιχειρήσεων. Μπορείτε να φανταστείτε ένα μοντέλο leasing, δηλαδή κάποιος να μην αγοράζει ε, κάποια προϊόντα, προϊόντα αλλά να τα νοικιάζει και να έχουμε μια κοινωνία παροχής υπηρεσιών και ο παραγωγός είναι και ιδιοκτήτης του προϊόντος και το ε, επανακτά μετά το τέλος της υπηρεσίας. Εσείς κάτι τέτοιο το υιοθετείτε, το υποστηρίζετε. Ευχαριστώ, συνάδελφοι, για τη συμπληρωματική ερώτηση. Το παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο στηρίζεται στην κατανάλωση και τη διασπάθηση πόρων. Ο κατασκευαστής κατασκευάζει κάτι χωρίς να νοιάζεται για τα απόβλητα πηγαίνει το προϊόν στον καταναλωτή και κάποια στιγμή θα πάει και αυτό στη χωματερή. Δεν γίνεται πια αυτό. Χρειάζεται νέο επιχειρηματικό μοντέλο, νέο οικονομικό μοντέλο, όπου ο κατασκευαστή, θα είναι υπεύθυνο για το προϊόν από την, από την κατασκευή του μέχρι την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωσή του. Υπάρχουν καινούργια σχέδια τώρα προϊόντων καινούριε ευθύνε για την επιστροφή των προϊόντων μέσα σε έναν κύκλο και πάνω σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ευχαριστώ πάλι κύριε Λάινεν. Η κυρία Κλάς, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πολλά μπορούμε να σκεφτούμε, πολλά να φανταστούμε, αλλά αυξάνεται ο παγκόσμιος πληθυσμός, ε, οι ενεργειακοί πόροι γίνονται όλο και πιο σπάνιοι και ο κόσμος πρέπει να αλλάξει. Πώς χειριζόμεθα τους σπάνιους αυτούς πόρους. Πρέπει να καλύψουμε όλο τον κύκλο ζωής ε, μεταφορά, μετατροπή, κατανάλωση, επαναχρησιμοποίηση και ε, από κομιδή. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά τους πόρους. Είναι σημαντικό και για την οικονομία και για την δημιουργία θέσεων εργασίας. Η επιμέρους πολιτική στόχη στην στρατηγική πρέπει να είναι όμως πολύ ε, Πολλές φορές ε, ε, ζητούμε αγρανάπαυση πολύτιμων ε, γεών ή τις απομονώνουμε. Αυτό γίνεται υπερβολη, με ο τρόπο. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μειώνουμε την παραγωγή τροφίμων σήμερα ιδίως. Νομίζω ότι στην Ευρώπη κάνουμε μεγάλη, δίνουμε μεγάλη συμβολή για την επίλυση των προβλημάτων του 21ου αιώνα. Ε, δηλαδή θέλουμε να καλύψουμε το πρόβλημα του επισητισμού, της κάλυψης με τρόφιμα ε, όλου του κόσμου προστατεύοντας παράλληλα τη βιοποικιλότητα. Η στρατηγική η ίδια θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην απέτηση ε, της αποτελεσματικότητας. Δεν μπορούμε δηλαδή να ε, ε, ψάχνουμε συνεχώς καινούργια μέτρα και κανόνες. Οι ισχύοντες κανόνες και οι ρυθμίσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται καλύτερα. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε και το ε, εργατικό δυναμικό ε, καλύτερα. Ε, οι υπερβολικοί δείκτες αυξάνουν τη γραφειοκρατία και σε τελευταία ανάλυση στοιχίζουν χρήμα και ενέργεια. Δεν είναι αποτελεσματικοί. Μην νομίζουμε ότι μπορούμε να ορίσουμε την αποτελεσματική διατροφή. Ε, μια καλή μπριζόλα νομίζω ότι είναι καλό τρόφιμο και ε, σηματοδοτεί καλή ποιότητα ζωής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τη συνάδελφε Κάντενμπαχ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η ECR είναι συντηρητική από μόνη της και δεν μπορούν να διατηρήσουν αυτό που μας είναι πολύ σημαντικό να συντηρήσουμε. Καθαρό αέρα, καθαρό νερό, καθαρό έδαφος. Το καταλαβαίνω. Δεν μπορούν να μας παρακολουθήσουν. Γιατί εμείς, άρα εμείς πρέπει να αναλάβουμε διπλή ευθύνη. Ευθύνη για την τωρινή γενιά, ευθύνη και για τις μελλοντικές γενιές. Αυτό θα το κάνουμε μόνο αν αντιμετωπίσουμε με περίσκεψη τις πρώτες ύλε και τους ενεργειακούς μας φόρους. Νομίζω ότι ο χάρτης πορείας εδώ ανοίγει πολλές δυνατότητες. Ε, όχι μόνο για τις οικονομικές επιδόσεις αλλά και για την αύξηση της ποιότητας ζωής. Δεν καταλαβαίνω αυτό το πανικό, αυτό το φόβο απέναντι στους φόρους τι είναι ο φόρο, Ο φόρος συμβάλλει στην ποιότητα ζωής. Τουλάχιστον στα γερμανικά ε, σημαίνει, ότι, ε, στα γερμανικά τουλάχιστον φόρο σημαίνει καθοδηγό επίσης ε, ετοιμολογικά. Ε, μπορούμε λοιπόν μέσα ε, από τους φόρους να καθοδηγήσουμε την Ευρώπη προς μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Είναι μέσα οι φόροι που μου επιτρέπουν να χρησιμοποιήσω τα χρήματα εκεί που χρειάζονται. Μιλήσαμε για την αρχή του ορυπαίνων πληρώνει. Ε, βέβαια, ε, οι φόροι θα πρέπει να είναι δίκαιοι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε απόψε τον κύριο Γκερμπράντι για την έκθεσή του και ελπίζω ότι θα, ε, γίνει, θα εγκριθεί με μεγάλη πλειοψηφία. Ευχαριστώ πολύ. Η συνάδελφη Γιόρνταν Ρωμάνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι Σήμερα ε, ε, οι άνεργοι στην Ευρώπη φτάνουν περίπου τα 24,8 εκατομμύρια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μια υγιή οικονομία. Η οικονομία ζητάει πόρους, ζητάει πρώτες ύλε και ε, άλλες συνθήκες που να επιτρέπουν τον ανταγωνισμό. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο φυσικό ρηκτό πλούτο, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο ε, φιδωλοί και αποτελεσματικοί στη χρήση των πόρων. Πώς θα γίνει αυτό. Δεν υπάρχει τρόπος να μας κάνει να τρώμε λιγότερο, να οδηγούμε λιγότερο, να αυξάνουμε τους φόρους συνεχώς. Δεν είναι αυτή η λύση. Η αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων και η εξοικονόμηση τους και των πρώτων υλών είναι η λύση. Αυτή είναι λοιπόν η ευκαιρία τώρα με νέο τρόπο λειτουργίας και της βιομηχανίας και της οικονομίας. Αυτό το έχει ξανασυζητήσει στο παρελθόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει μάλιστα εγκρίνει και αντίστοιχη γνωμοδότηση μετά από μήνες συζητήσεων. Δεν είναι μέτρα λιτότητας αυτά που συζητούμε. Είναι ένα θέμα που δεν απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης, ε, ε, αλλά δεν χρειαζόμαστε νέα μέτρα ούτε ε, νέα σύμφωνα. Ε, αρκούν αυτά που έχουμε, αλλά θα πρέπει να τα υλοποιούμε, να τα εφαρμόζουμε σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τις κατευθυντήριες γραμμές. Και θα πρέπει να έχουμε και ένα πολυετή ε, προπολογισμό. Δεν θα πρέπει να λέμε στον κόσμο ότι ο μικρός προπολογισμό είναι ο καλός προπολογισμό. Να είναι ο σωστός προπολογισμό. Αυτό μα ενδιαφέρει. Ε, ο προπολογισμό που χρειάζεται κάθε φορά για να εφαρμόζεται η νομοθετία. Έχουμε δείκτες που μας βοηθούν να μετρούμε την ε, εξοικονόμηση πόρων και την αποτελεσματική χρήση. Παρακαλώ, συνεχίστε κύριε Επίτροπε. Τώρα ο κύριο Τανασέσκου, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι. Έχουμε μεγάλες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε σήμερα στην κοινωνία μας. Και δεν είναι εύκολη η απάντηση ούτε να δοθεί ούτε να βρεθεί για την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον εισηγητή και τους και εισηγητές για το έργο τους. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι ότι γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, γνωρίζουμε προς τα πού θέλουμε να πάμε και το μόνο που ε, μας μένει είναι να ακολουθήσουμε τους στόχους μας για να τους υλοποιήσουμε. Πολλά θα πρέπει να γίνουν σε τοπικό επίπεδο ή περιφερειακό αρκεί να σκεφτώ την επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων ε, των αστικών αποβλήτων, ας πούμε. Υπάρχουν χώρες ε, όπου έχουν καταργηθεί τελείως ηχητά όπω όπως η Γερμανία και οι κάτω χώρες, αλλά υπάρχουν και άλλες ε, ε, χώρες που έχουν ακόμα μεγάλες χωματερές. Και σε αυτές ανήκει και η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Το Βέλιο και η Σουηδία είναι κάπου στα μισά του δρόμου, αλλά στη σωστή κατεύθυνση τις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης στην Ρουμανία είναι ε, και ε, η έγκριση μιας εθνικής στρατηγικής για την ανακύκλωση των αποβλήτων οι ε, κρατικές αρχές και οι τοπικές και οι περιφερειακές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και για την αποδοχή της ευρωπαϊκής ατζέντα. Ε, αλλά ε, όχι μόνο γι' αυτό, γιατί αυτές καλούνται να υλοποιήσουν στη συνέχεια τις στρατηγικές αυτές. Θα πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν τι συμβαίνει και να τους έχουμε στο πλευρό μας. Όλο και περισσότεροι πολίτες πιστεύουν στην αηφόρο κατανάλωση και αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε κι εμείς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πέτερλε. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έδωσε μια καλή βάση για να κάνουμε μια καλή έκθεση. Και θα ήθελα να συγχαρώ και τον εισηγητή και την Επιτροπή. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στην αηφόρο ανάπτυξη χωρίς ε, σωστή αξιοποίηση των πόρων. Καλωσορίζω την ε, πρόταση, τη συνολική, ε, που έχονται όλοι και οι νομοθέτες και η παραγωγή και η βιομηχανία και η κοινωνία των πολιτών. Χαίρομαι γι' αυτό. Επίσης, ε, χαίρομαι για το νέο σύστημα δικτών που προτείνεται. Είναι ο μόνος τρόπος ακριβώς να μετρήσουμε την πρόοδο που επιτελούμε. Επίσης, υποστηρίζω την πρόθεση να συμπεριληφθεί αυτή η προσπάθεια και στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Υποστηρίζω την έκκληση να καταργηθούν όλες οι επιδοτήσεις ε, σε ρηπογόνους κλάδους. Είναι υπεύθυνη η στάση αυτή επέναντι στην Ευρώπη, αλλά ε, και θα βοηθήσει να αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες, νέες θέσεις απασχόλησης. Επίσης υποστηρίζω την καλύτερη λειτουργία ε, της αγοράς ανακύκλωσης στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τις ζωικές πρωτεΐνες, το θέμα δεν είναι ε, μόνο να αξιοποιούμε καλύτερα ε, την υπεθρό, αλλά βοηθάει και στην υγεία μας αυτό. Ευχαριστώ κύριο Περέλο Ροντρίγκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ενώ ποιό μας έχουμε μια έκθεση του κυρίου Γκερμπράντη, τον οποίο θέλω να συγχαρώ κατά τα άλλα, που μαζί με τον οδικό χάρτη είναι τα δύο καλύτερα παραδείγματα που μας δείχνουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε και που θέλουμε να ακολουθήσουμε από το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά ο, καμί... ο δρόμος αυτός είναι στρωμένος και με εμπόδια. Κρίση, λιτότητα λέγονται αυτά, καμιά φορά λέγονται και επικουρικότητα που χρησιμοποιείται ως εμπόδιο και ε, άλλες φορές μας λέγουν ότι δεν είναι εφικτά. Φτάνει πια. Θα πρέπει να ε, διδαχθούμε από τα σφάλματά μας, όχι πια εμπόδια. Για να έχουμε μια υφόρο ανάπτυξη θα πρέπει να αξιοποιούμε καλύτερα τους πόρους, να τους χρησιμοποιούμε καλύτερα και να μην ε, τους σπαταλούμε με τον τρόπο που κάνουμε μέχρι σήμερα. Γι' αυτό θα ζητούσα από τον Επίτροπο να μας πει. Ποια θα είναι τα μέτρα εκείνα που πρέπει να εφαρμόσουμε, τα διορθωτικά για να μην έχουμε αύξηση των τιμών λόγω της σπάνης ε, των πόρων. Να έχουμε ε, χαμηλό ΦΠΑ για τις δευτερογενείς ύλες, για να μπορούμε να ανακυκλώνουμε περισσότερο. Θα πρέπει ε, να μετακινηθεί και η φορολογία από τη φορολόγηση της εργασίας στη φορολόγηση των κερδοσκοπικών κινήσεων κεφαλαίων. Ουσιαστικά ζητούμε δέσμευση, απέτηση, γιατί υπάρχουν χώρες που μειώνουν ε, τις ε, δαπάνες για την έρευνα, για την παιδεία, για την υγεία, όπως η δική μου χώρα και δεν είναι στο σωστό δρόμο. Απαιτήστε περισσότερα από εκείνους, παρακαλώ. Κύριο Σκέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πιο σημαντικό θέμα είναι να παραμείνει η Ευρώπη οικονομικά ανταγωνιστική για το μέλλον. Πράγμα που θα βελτιώνει τι ε, συνθήκε διαβίωση των συμπολιτών μα και θα μα κάνει πιο ανεξάρτητου αυτή τη στιγμή είμαστε εξαρτημένοι από τους σπόρους και πρέπει να δούμε τι έχουμε οι ίδιοι και να το αναπτύξουμε. Καταρχήν να μειώσουμε τα οικιακά απόβλητα και το τεράστιο όγκο τους. Πρέπει πληρούνται οι συνθήκες για να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Τα παιδιά όταν περνάνε από το δημοτικό στο γυμνάσιο ε, έχουν ε, βαθμολογία όσον αφορά την στάση τους προς το περιβάλλον. Είναι σημεούλα. Ε, πραγματικά είναι κατάλληλη στιγμή για να βελτιωθούμε προς αυτό το τομέα. Ε, η γεωργία είναι ένα τεράστιο τομέα, Πρέπει να εξασφαλίσουμε ασφάλεια των τροφίμων και ταυτόχρονα το ότι όλα γίνονται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Η ενέργεια φυσικά είναι πολύ σημαντική και ε, ενώ έχουμε κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά την ε, ενέργεια και ιδιαίτερα τον άνθρακα γιατί μολύνει, ρηπαίνει πολύ θα πρέπει να μιλήσουμε και για το φυσικό αέριο από σχιστόλιθο και ε, όλα τα, όλες τις δυνατότητες που έχουμε για να αναπτυχθούμε στο μέλλον και εδώ έτσι έρχομαι στη σημασία της έρευνας. Το Horizon 2020 που μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε έρευνα σε αυτούς τους τομείς, να χρησιμοποιήσουμε τους φυσικούς πόρους που έχουμε. Και τέλος θέλω να αναφέρω την μπλε οικονομία. Πριν από λίγε εβδομάδε είχαμε μια επίδειξη στι Βρυξέλλες που περιέγραφε το ευρύ ε, δυναμικό που προσφέρει η θάλασσα όσον αφορά τα τρόφιμα, τις ε, τροφές και άλλους τομείς ε, επίσης. Ε, σας ευχαριστώ. Ο κύριος Αρσένης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πραγματικά, Επίτροπε, ο τεράστιο αριθμό ομιλητών στη σημερινή συζήτηση δείχνει το πώ το Κοινοβούλιο στηρίζει την πρωτοβουλία σα και πραγματικά ενδιαφέρει να προχωρήσουν προ αυτή την κατεύθυνση. Και είναι λογικό γιατί 16 τόνου ε, υλικών καταναλώνει χρησιμοποιεί ε, κατά μέσο όρο ένας ε, ευρωπαίος πολίτης. έξι τόνοι από αυτού πάνε στα σκουπίδια. το κόστος είναι τεράστιο. καταλαβαίνω ότι πολλοί συνάδελφοι αντιδρούν σε αυτές τις ιδέε, όμως δεν καταλαβαίνω το γιατί. έχουμε μια οικονομική κρίση τεράστια απέναντί μας και δεν είναι μόνο με τη μείωση των δεν είναι μάλλον καθόλου με τη μείωση των χαμηλών μισθών και συντάξεων που θα τη λύσουμε. Πρέπει να σταματήσουμε την εισαγωγή προϊόντων και υλικών που καταλήγουν στα σκουπίδια μα. Γι' αυτό, Επίτροπε, προχωρήστε στην πρωτοβουλία σα αυτή και παρακαλώ προχωρήστε ακόμα πιο δυναμικά με δεσμευτικού στόχου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αν το σύστημά μας είναι να καταρρεύσει, ε, το, τον οικονομικό μας σύστημα καταρρεύσει, μπορούμε να βρούμε τρόπο να, να τη γλιτώσουμε. Όμως αν καταρρεύσει το σύστημα των πόρων μας, τότε πάει τέρμα. Ε, το παιχνίδι τελειώνει. Ε, και προς τα εκεί κατευθυνόμαστε και γι' αυτό νομίζω πως είναι μια καλή αρχή αυτή η έκθεση, αλλά σίγουρα πρέπει και να προχωρήσουμε. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένους ορισμούς για τους πόρους, για τα οικοσυστήματα, για καλύτερη χρήση της, ε, των πόρων χρειαζόμαστε δείκτες τόσο για τους προϋπολογισμούς μας όσο και σε ε, εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό πρέπει να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στοιχεία στη στρατηγική ανάπτυξη ε, και στο ευρωπαϊκό εξάμενο και χρειάζεται μια αποτελεσματική οδηγία οικολογικά σχεδιασμένη με συγκεκριμένους δείκτες για την δυνατότητα ανακύκλωσης ε, κάθε προϊόντος και θα ρίνω την Κομισιόν να δράσει σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σταμπάιτζη. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε πραγματικά ένα καλό σχέδιο γιατί θέλουμε ε, πραγματικά μια οικονομία που να ε, αξιοποιεί τους πόρους και να διαχειρίζεται σωστά τα απόβλητα. Το 2012 μεταξύ άλλων είναι και το έτος που προσφέρεται ε, για αυτές τις προσπάθειες. Αν συγκριθούμε με άλλες χώρες του κόσμου, διαπιστώνουμε ότι το Ισραήλ Φερρυπίν έχει κάνει πολύ περισσότερα από εμάς. Εκεί έχουν λειψιδρία και είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε και εμείς αργότερα. Τώρα, το θέμα της ανακύκλωσης, της επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων ε, είναι επίσης πολύ σημαντικό. Δυστυχώς, στην Ουγγαρία, τη χώρα μου, Πολλά είναι ακόμα στρεβλά και χαμηλές οι επιδόσεις που έχουμε εμείς να επιδείξουμε. Είναι καλό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα δεσμευτικό σύστημα. Μαζέη Κοκοβίτς. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, και κύριε Ισηγητά. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά και εσείς προσωπικά κάνατε πάρα πολλά. Φανταστείτε την Ευρώπη ως ένα ασθενή που πάσχει από μία χρόνια νόσο και θα πρέπει να αλλάξει τελείως τον τρόπο ζωής της. Μερικοί το κάνουν αυτό και μακροβιούν και είναι υγιείς και ε, δεν έχουν προβλήματα. Οι άλλοι όμως που δεν μπορούν να προσαρμοστούν συνεχίζουν τον παλιό τρόπο και στυλ ζωής και πεθαίνουν από την ασθένεια αυτή. Γι' αυτό θα πρέπει λοιπόν και στην Ευρώπη να αυξήσουμε την ανάπτυξη, την απασχόληση και να χρησιμοποιούμε καλύτερα τους πόρους. σε καιρού κρίση είναι πιο εύκολο να γίνει αυτό ε, σε εποχές παχιών αγελάδων. Είναι γεγονός ιστορικό ότι η αυθονία δεν βοηθάει στην εφευρετικότητα και τη δημιουργικότητα. Οι πολίτες μας θα μπορούσαν ε, πραγματικά να κάνουν πολλά εάν τους εξηγούσαμε με ποιο τρόπο πρέπει να λειτουργήσουμε. Είναι η καλύτερη ευκαιρία να πετύχει η πολιτική και να συμμετέχει ολόκληρη η κοινωνία. Έχει ανοίξει η πόρτα για την έρευνα, για την καινοτομία και η Ευρώπη είναι ένας πολύ ωραίος τόπος ε, για έρευνα, για δημιουργικότητα, για εφευρέσεις. Έχουμε δίκτυα, έχουμε καλές αγορές και όλοι θα πρέπει να εξοικονομούμε πόρους για να μην εξαρτώμαστε τόσο πολύ από τρίτες χώρες και να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης. Ο κύριος Σόνικ. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η οικονομία μας ε, αντιμετωπίζει κρίση και οι περιβαλλοντικοί πόροι μειώνονται ε, και η Ευρώπη θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, να εγγυηθεί την αδιάκοπτη ανεφοδιασμό σε πόρους. Ε, θα πρέπει επίσης να πιο λογικά να χρησιμοποιεί και πιο αποτελεσματικά τους πόρους έτσι ώστε να προστατευτεί το περιβάλλον αλλά και να αποτεμιευθούν πόροι. Θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα χρησιμοποιώντας και καταναλώνοντας λιγότερα. Δεν μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε να ακολουθούμε το ίδιο πρότυπο. Πρέπει να κοιτάμε την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Αυτό είναι θέμα κλειδί και όσον αφορά την εγγύηση για την οικονομική ανάπτυξη και για την απασχόληση εδώ έχουμε να κάνουμε με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των πόρων, νέες δυνατότητες, θα πρέπει να εγγυηθούμε αυτές τις ιδέες χωρίς να βλάψουμε την ανταγωνιστικότητά μας Μιλάμε για την απασχόληση, για την τεχνολογική ανάπτυξη, για την ανάπτυξη των πράσινων τεχνολογιών και τη διατήρηση των διαφόρων οικονομικών ε, πτυχών στην Ευρώπη. Αυτό το φιλόδοξο σχέδιο δεν αρκεί μόνο του. Ε, είμαι ευτυχής που έχει ως στόχο ο κ. Ζουκερμπράντι να περιορίσει και τη γραφειοκρατία. Ε, θέλουμε να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά οι κείμενες νομοθεσίες και να χρησιμοποιήσουμε για όλα τα κρατημέλη, μάλλον να ορίσουμε για όλα τα κρατημέλη ρεαλιστικούς στόχους, γιατί εάν όχι η στρατηγική μας δεν θα έχει ε, χρησιμότητα. Το μέλλον μας εξαρτάται από το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τους πόρους τώρα. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να έχουμε μια ισορροπημένη στρατηγική. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Η κυρία Μπασέσκου καταρχήν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για να υπερβούμε τη σημερινή οικονομική κρίση, καλούμαστε να βρούμε νέες μεθόδους ε, για την ανάπτυξη, ε, ένα φιλόδοξο σχέδιο για τη μελλοντική μας ανάπτυξη. Θα πρέπει να αυξήσουμε και το επίπεδο το βιωτικό και την ευημερία μας. Η οικονομική απόδοση όμως σημαίνει ε, και ορθολογική χρήση των πόρων, γιατί οι πόροι είναι πεπερασμένοι. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι τα ορυκτά δεν αναπαράγονται Ούτε το έδαφος, ε, ούτε ε, ο ατμοσφαιρικός αέρας, ούτε το νερό είναι ανεξάντλητα. Ήδη καταναλώνουμε περισσότερα από όσο ε, μπορεί να παράγει η γη. Και ιδιαίτερα στην Ευρώπη είναι πολύ ψηλή κατανάλωση. Γι' αυτό χρειάζεται ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση και προγράμματα ενημέρωσης για να αλλάξουν οι συμπεριφορές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Γιασροβιέσκα. Στο παρελθόν, τα τελευταία χρόνια γνωρίσαμε μεγάλες κρίσεις και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ε, υπάρχει ε, πρόβλημα, ε, οι πόροι είναι πεπερασμένοι ε, και τα ορυκτά. Ας πούμε, τα σπάνια ορυκτά είναι κάτι το οποίο στο μέλλον θα παίξει μεγάλη σημασία και αυτά δεν βρίσκονται στην Ευρώπη. δεν θα πρέπει να δημιουργούμε ε, συνεχώς νέα όργανα που να συζητούν στρατηγικές οι οποίες δεν θα εφαρμόζονται. Χρειάζονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, συγκεκριμένα έργα και σχέδια. Είμαι πεπισμένη ότι αυτές οι πρωτοβουλίες και αυτά τα σχέδια ε, θα μπορέσουν να μας οδηγήσουν στο στόχο. Αν θέλουμε και μπορούμε να χρησιμοποιούμε τους πόρους αποτελεσματικά, όχι, ε, ε, δεν θα είμαστε μόνο ανεξάρτητοι από εκείνους που έχουν σήμερα το ρηκτά, αλλά θα διαφυλάξουμε και τις θέσεις ε, εργασίας. Ευχαριστώ, κυρία Μπιλμπάου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεση για την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Τονίζω την ιδέα των μονίμων υλικών σε σχέση με τις πρώτες ύλες που ε, είναι πεπερασμένες. Θα πρέπει να βοηθάμε και τους παραγωγούς και τους χρήστες και τους καταναλωτές ε, για να ανακυκλώνονται τα υλικά. Για τα απόβλητα έχουμε στόχο μείωση της παραγωγής αλλά και καλύτερης ε, ανάκτησης και ανακύκλωσης. Οι στόχοι μας θα πρέπει να είναι βιώσιμοι, ρεαλιστικοί, να χρησιμοποιούμε καλύτερα αυτά που ανακυκλώνονται και καλύτερα να διατίθενται τα μη ανακυκλώσιμα απόρριτα. Θα πρέπει να στηρίζουμε τεχνολογίες καινοτόμες ε, για την ανακύκλωση των αποβλήτων. Θα πρέπει να ε, τερματιστούν οι χώροι γενομικής ε, ταφής αποβλήτων και τα μη ανακυκλώσιμα απόβλητα να αποτεφρώνονται. Χρειάζονται περισσότερε απαιτήσει από τα κράτη-μέλη και τι περιφερειε. Η πρόκληση μα αφορά όλου και θα πρέπει όλοι να συμμετέχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, οι βιομηχανοποιημένες ε, κοινωνίες ε, δέχονται μεγάλες επιθέσεις όσον αφορά τις ε, μεγάλες πιέσεις όσον αφορά τους ολοένα και πιο σπάνιους και λιγοστούς πόρους. Θα πρέπει λοιπόν ε, να σεβαστούμε και να προστατεύσουμε το κοινό συμφέρον και για τις μελλοντικέ γενναίες. Ο περιορισμός της κατανάλωσης και ανακύκλωση καθώς και η αποτελεσματική χρήση των πόρων είναι επιτακτικές ανάγκες, αλλά δεν πρέπει αυτό να αφαιθεί στις, ε, στη βούληση της αγοράς, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι. βιώσιμοι και αποτελεσματική χρήση των πόρων απαιτεί βαθιά αλλαγή των μοντέλων παραγωγής και κατανάλωσης που ισχύουν. Για παράδειγμα, θα πρέπει να αμφισβητήσουμε το ελεύθερο εμπόριο και την χρήση της ενέργειας που αυτό σημαίνει. Ε, τις ε, σύντομες αλυσίδες ε, ανεφοδιασμού. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε να βάψουμε πράσινο ένα σύστημα που έφτασε σε αυτή την κοινωνία σε... και να τις κάνει το βίο αβίωτο. Ευχαριστώ. Ακόμα και οι όσοι αφισβητούν τις κλιματικές αλλαγές θα πρέπει να σκεφτούν ότι οι πόροι είναι ε, πέρατη και ε, βεβαίως ε, αυτοί που δεν, που δεν τελειώνει ο πόρος είναι η ποιότητα των λαών μας. Αν δούμε την σελίδα 7 του εγγράφου του 2010 της Κομισιόν Ευρώπη 2020 λέει πω η Ευρώπη έχει πολλές δυνάμεις και μπορούμε να βασιστούμε στο ταλέντο και τη δημιουργικότητα των λαών μας. Σπάνια παραδοχή αυτή κάποιο κουμπί θα ξεχάσαν να πατήσουν. Συνήθως ε, ε, τα ιδεολογικά εγκλήματα δεν επιτρέπονται. Όμως είχε δίκιο η Κομισιόν. Τα επιτεύγματα των λαών της Ευρώπης ε, στις, στη τεχνολογία και στις τέχνες είναι άνευ προηγουμένου. Γιατί όμως είμαστε τόσο αργοί και γιατί θέλουμε να αντικαταστήσουμε τους λαούς της Ευρώπης με λαούς από άλλα μέρη του κόσμου που ήταν λιγότερο τυχεροί όσον αφορά τη... Ευχαριστώ. Κυρία Μαγκίνας, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή. Παλιότερα λέγαμε ότι δεν πρέπει να ε, σπαταλάμε, δεν πρέπει να θέλουμε. Μετά προσπαθήσαμε να εξευγενήσουμε λίγο αυτή την προσέγγιση και να την κάνουμε πιο φιλική προς τον κόσμο. Διαβάζοντας ε, μέρη της έκθεσης, βλέπω ότι μάλλον παραλύει, παρακινητοποιεί. Δέχομαι ότι έχετε καλές προθέσεις. Ιδιαίτερα στις διατροφικές συνήθειες πρέπει να αλλάξουν, στη χρήση της γης πρέπει να αλλάξει και συμφωνώ με την παράγραφο 56 σε σχέση με τη χρήση γης ε, και τι πρέπει να παράγουμε. Θα πρέπει όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παράγουμε περισσότερους πόρους. Επίσης η παράγραφος 57 είναι πολύ καλή γιατί βελτιώνει την ενημέρωση του καταναλωτή. Η 58 όχι τόσο. Νομίζω ότι καλύτερα θα ήταν να χρησιμοποιούμε λιγότερα λόγια ε, όπως το, στους προηγούμενους αιώνες ε, και να καταλήξουμε στο ίδιο. Μην ε, σπαταλούμε, μην ε, ζητάμε πολλά. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Ματούλα. Ευχαριστώ πολύ. Καλύτερη, αποτελεσματικότερη χρήση πόρων, αποτελεσματική χρήση ενέργειας. Και τα δύο είναι σημαντικά για διαρκή και βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2020 και μετά. Την επόμενη δεκαετία οι ανανεώσιμες ενέργειες ως ε, ποσοστό θα αυξηθεί. Ε, υπάρχουν όμως διαφορετικές δυνατότητες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το φυσικό αέριο στο μέλλον, στο ενεργειακό μείγμα της Ένωσης, θα έχει τη σημασία του, υπό την προϋπόθεση ότι και οι νέες μορφές αξιοποίησης του αερίου θα αξιοποιηθούν, ε, θα λυθούν υπόψη. Επίσης, να λάβουμε υπόψη μας ότι καμιά φορά χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις ώστε η ενέργεια να μεταφερθεί από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Όμως ε, εδώ θα μπορούσαμε να εντάξουμε και ιδιώτες επενδυτές. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά, λέει ο κ. Μικολάσικ. Αν συνεχίσουμε έτσι, αν αξιοποιούμε, χρησιμοποιούμε αναποτελεσματικά τους πόρους μας, θα έχουμε κακό τέλος. Ε, ιδιαίτερα θα πληγούν ε, τα πιο φτωχά στρώματα του πληθυσμού. Όλοι γνωρίζουν ότι η Ευρώπη έχει λιγότερους σπόρους, άρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους σπόρους αυτούς αποτελεσματικότερα. Η οικονομική κρίση έχει ως συνέπεια να επιδιώκει η Ευρώπη αναγκαστικά νέες δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης. Ε, θα πρέπει να συνδυαστούν αποτελεσματικότερα οικονομική και κοινωνική πολιτική. Χρειάζονται οράματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο τελευταίος ομιλητής είναι ο κύριος Λουβάν, από ό,τι βλέπω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρώπη είναι αποτελεσματική στην χρήση των πόρων της. Χρειαζόμαστε όμως καινούρια μοντέλα καταναλωτικής συμπεριφοράς και καινούρια διακυβέρνηση στον τομέα της καταναλωτικής συμπεριφοράς όλο το ενεργειακό τοπίο της Ευρώπης πρέπει να αναδιαρθρωθεί. Θα πρέπει και σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο να υπάρχει συμμετοχή και ενδιαφέρον για την καινούργια αυτή προσέγγιση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει υποχρεωτικούς δεσμευτικούς στόχους που θα καλύπτουν δημοκρατικές συμβάσεις στην ενέργεια και τις ενεργειακές υποδομές και αυτό ως μέρος της στρατηγικής που πρέπει να ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια η Ευρώπη. Και υπάρχει, ε, υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Όχι. Παρακαλώ, Επίτροπε Ποτότσνικ. Έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν πρέπει να πω ότι αυτή ήταν η πρώτη πραγματική ολομέλεια στην οποία συμμετείχα και αυτό το εκτιμώ όλος ιδιαιτέρως, ε, είναι μεγάλη ενθάρρυνση. Προκειμένου να απαντήσω στα πολλά που είπατε, από τη γενοτομία, τη γεωργία, την αλληλεία, τους δείκτες, τους στόχους, την ολοκλήρωση, ε, διατροφικές αλλαγές κλπ. Σχεδιασμός νέων τροφίμων. Α, αν επρόκειτο να τα κάνω όλα αυτά θα χρειαζόμουν πολύ χρόνο. Είναι δε και σύνθετα τα θέματα που συζητούμε. Και καμιά φορά δεν είναι τόσο εύκολο να απαντήσει κανείς αλλά ως ε, Επίτροπο Περιβάλλοντος θα επικεντρωθώ σε κάποιες ανησυχίε που εξέφρασαν ορισμένοι συνάδελφοί σα, εδώ που αφορούν το θέμα της οικονομίας και την σημερινή κατάσταση και γιατί αυτά που αναφέρονται στην έκθεση Gerbrand είναι τόσο σημαντικό να υποστηριχθούν. Αρχίζω με τον 20ο αιώνα που ήταν ε, ένα μοντέλο εντατικής χρήσης των πόρων αυξήθηκε τέσσερις φορές ο πληθυσμός, η οικονομική παραγωγή αυξήθηκε στο πολλαπλάσιο και οι πόροι αυξήθηκαν αντιστοίχως. Εκείνη την, στη χρήση τους. Η τιμή των πόρων με τον ε, σύνθετο δίκτυ ε, ε, μειωνόταν και δεν υπήρχε η σκέψη ότι ήταν περασμένη στο μοντέλο που χρησιμοποιούσαμε. Αυτό αλλάζει γιατί αυξάνεται ο πληθυσμός, θα φτάσουμε στα 9 δις το 2050, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι το 2030 αναμένουμε 3 δις ανθρώπων που θα περάσουν από το επίπεδο της φτώχειας στο επίπεδο των μεσαίων στρωμάτων που όμως δεν θα μπορούν να ζήσουν ως μεσαία στρώματα αν συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε το μοντέλο που είχαμε τον 20ο αιώνα. Τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη. Η Ευρώπη ε, ε, ε, έχει πολλές εξαρτήσεις. Οι τιμές πολλών πόρων την τελευταία δεκαετία αυξάνονται πλέον και αυτό είναι μια τάση που αναμένεται από τις περισσότερες εταιρείες το 85% και οι διακυμάνσεις αυτών των τιμών είναι τεράστια. Σήμερα λοιπόν ο ευρωπαϊκός επιχειρηματικός τομέας επαναστοχεύει ε, την παραγωγικότητα της εργασίας, στην παραγωγικότητα των πόρων, γιατί βλέπει ότι εκεί βρίσκεται η μεγάλη πρόκληση και οι μεγάλες ευκαιρίες. Παραγωγικότητα σε σχέση με τους πόρους, όχι πια τόσο πολύ παραγωγικότητα εργασίας. Λοιπόν, ε, ε, υπάρχουν πάρα πολλοί πόροι που είναι κρίσιμοι, κέρια σημασίας. Καμιά φορά ε, ε, έχουμε το νερό, έχουμε τη γη που είναι πεπερασμένη πόροι και είναι αντικείμενο μεγάλης προσοχής. Η φύση δεν έχει μπει τόσο πολύ μέσα στο τοπίο αυτό, αλλά θα γίνει αυτό. Αυτές είναι οι νέες προκλήσεις. Τώρα πώς συνδέονται όλα αυτά με την κρίση που ζούμε όλοι, ε, την ανάγκη για ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Όπως είπε ο Όλι Ρέν στην ομιλία του πριν από μια μέρα, αν είχαμε μια σημαίνια σφαίρα, θα την είχαμε ήδη χρησιμοποιήσει, αλλά δεν την έχουμε. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να δουλεύουμε υπομονητικά, αργά, ε, αξιοποιώντας τους, το, τους δυνατούς τομείς μας όπως το ταλέντο, η οικονομία της γνώσης, η έρευνα, η καινοτομία. Ένας άλλος ε, τομέας είναι η απόλυτη επάρκεια πόρων. Αν χρησιμοποιούμε λιγότερο νερό, λιγότερη ενέργεια, λιγότερες πρώτες ύλες, αν παράγουμε ανακυκλώσιμα προϊόντα, αυτό έχει νόημα ε, ε, με οικονομικούς όρους. Και αυτή είναι μια τάση η οποία όλο και περισσότερο χαρακτηρίζει τις επιχειρήσεις και την οικονομία. Μιλάμε λοιπόν για οικονομική και περιβαλλοντική ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα ταυτόχρονα και προσεγγίζουμε ταυτόχρονα τα δύο θέματα. Έτσι λοιπόν, κατανοώ τον κατεπήγοντα χαρακτήρα της εφαρμογής των μέτρων. Αυτό είναι το σημαντικό και προσπαθούμε να επιστήσουμε την προσοχή σε αυτό και όταν μιλάμε για το, ε, την ιστορία των εξαμήνων και το κέντρο της οικονομικής διακυβέρνησης και συζητούμε για όλα αυτά τα θέματα τα οποία οδηγούν στην καλή χρήση των πόρων. Ε, ένας συνάδελφός σας είπε πολύ σωστά ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε τους φόρους. Ε, δεν ε, προτείνουμε τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο από το να περάσουν οι φόροι από την εργασία που έφτασαν πολύ ψηλά, έχουμε υψηλό εργατικό κόστος. Μετατόπιση των φόρων από την εργασία λοιπόν στους πόρους. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να μειώσουμε τους επιβλαβείς ε, πόρους ε, αλλά και τις επιδοτήσεις όταν ε, ψάχνουμε να χρησιμοποιήσουμε και τα κονδύλια που διαθέτουμε με καλύτερο τρόπο. Είναι σημαντικό λοιπόν να συμβουλέψουμε τα κράτη-μέλη που έχουν την ευθύνη να πάρουν αυτά τα μέτρα. Και ήδη το Μάρτιο του 2011 στα συμπεράσματα ε, είχαν υποστηριχθεί οι προτάσεις αυτές. Επίσης εργαζόμεθα πολύ για την εφαρμογή του χάρτη πορείας, του roadmap που φέτος θα εστιαστεί πολύ στο νερό. Θα αρχίσω με, με την πλατφόρμα μεταβίβασης ε, στην αποτελεσματικότητα των πόρων σε λίγες μέρες, πράγμα που θα δώσει ορμή και όθηση θα είναι κομμάτι του προγράμματος για το περιβάλλον όπως πρέπει άλλωστε και Βέβαια, ο κατεπήγον χαρακτήρας της εφαρμογής είναι στην καρδιά του προβλήματος. Θα το συζητήσουμε σε λίγες μέρες στο Ρίο συνήκωση στη Σύνοδο Κορυφή. Δεν θα μιλήσω για την αποτελεσματικότητα των πόρων, αλλά για την πράσινη οικονομία. Αλλά το ίδιο πράγμα είναι. Ούτε θα μιλήσουμε μόνο για την Ευρώπη, αλλά για συνολικέ δεσμεύσει. Γιατί Όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτά είναι τα πραγματικά αναγκαία πράγματα. Τέλος, αν όλα πήγαιναν καλά με την καφέ οικονομία και την ανάπτυξη, δεν θα μιλούσαμε για την πράσινη τώρα. Όμω η καφέ ανάπτυξη και βιομηχανία έχει όρια στην ανάπτυξη που αναγνωρίζονται σήμερα από τον επιχειρηματικό τομέα. Πρέπει και εμεί οι πολιτικοί να αναγνωρίσουμε τα όρια αυτά. Και όταν μιλάμε για την πράσινη ανάπτυξη, μιλάμε για το πώς θα σχεδιάσουμε την ανάπτυξη του μέλλοντος που θα οδηγήσει σε ευμάρεια και ωφέλη περισσότερα από ό,τι φέρνει αυτή τη στιγμή η καφέ οικονομία. Δεν θέλω να καταστροφολογώ γιατί είμαστε ε, ευφυείς κοινωνίες, είμαστε, είναι ευφυές το ανθρώπινο είδος. Όμως ε, το βιο, ε, το, το αηφόρο μέλλον, η βιωσιμότητα ε, δεν είναι επιλογή, είναι ε, ανάγκη, είναι ένα δεδομένο. Σας ευχαριστώ όλους όσους μείνατε μέχρι το τέλος της συζήτησης. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τη δευτερολογία σας και τον τελικό λόγο έχει τώρα ο συγκητής μας ο κύριος Κερμπράντη. Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να αρχίσω με ευχαριστίες προς τους συναδέλφους μου για την ευρύτατη υποστήριξη που γνώρισε η έκθεσή μου. Μου κάνει πάρα πολύ καλό. Άκουσα πολύ προσεκτικά και διαπίστωσα πολύ μεγάλη συνένεση για τον τελικό στόχο, την πιο αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Μπορεί να διαφωνούμε για το δρόμο που θέλουμε να ακολουθήσουμε και για τους ρυθμούς με τους οποίους θα προχωρήσουμε. Θέλω όμως να πω το εξής. Η ταχύτητα που μπορούμε να επιτρέψουμε σε αυτούς μας δεν είναι κάτι που επιβάλλουμε εμείς η Ευρώπη, αλλά το επιβάλλει ο κόσμος σε μας. Και είναι τόσο μεγάλη η ταχύτητα αυτή που δεν μπορούμε να μην έχουμε φιλόδοξους στόχους και φιλόδοξη ατζέντα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκφράστηκε κάποια κριτική για τον οικολογικό σχεδιασμό Επιτρέψτε μου να πω το εξή: Το κείμενο αυτό που συζητούμε σήμερα δεν είναι νομοθετικό και που ψηφίζουμε αύριο. Είναι πολιτικού περιεχομένου, όχι νομοθετικού περιεχομένου. Δείχνει τη βασική κατεύθυνση για την πολιτική του μέλλοντος. Δηλαδή δεν μπαίνει σε λεπτομέρειες για το πώς ε, θα πρέπει να, να προσαρμοστεί η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό. αλλά όταν ε, φτιάχνουμε κάποια προϊόντα από το σχεδιασμό τους ήδη θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι πρώτες ύλε πρέπει να επανακτηθούν και να χρησιμοποιηθούν. Πρόεδρε, το σημαντικότερο της έκθεσης αυτής είναι ότι ως Κοινοβούλιο θα στείλουμε ένα πολύ χειρό και στεναρό πολιτικό μήνυμα και θα υποστηρίξουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προχωρήσει στο δρόμο που χάραξε. Και όχι μόνο να προχωρήσει, αλλά να ε, δείξει και πολύ μεγαλύτερη φιλοδοξία από τη σήμερα στην ατζέντα και στο πρόγραμμά της. Και αυτό έχει να κάνει με την εφαρμογή και με την νομοθεσία τώρα. Στη σημερινή συζήτηση Ορισμένοι θεώρησαν ότι είναι διαζευτικό αυτό ή το ένα ή το άλλο. Όχι, είναι και το ένα και το άλλο. Και πρόεδρε, θέλω να πω και κάτι για το Συμβούλιο. Ασταλεί ένα μήνυμα πολύ ηχηρό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα κράτη-μέλη ότι έχουμε φιλόδοξο πρόγραμμα και θέλουμε να προχωρήσουμε. Όχι μόνο γιατί μας αρέσουν εμάς όλα αυτά, αλλά γιατί είναι επίγουσα ανάγκη για την ευρωπαϊκή οικονομία. Όπως δεν περίμεναν οι χρηματαγορές να είναι έτοιμοι οι ηγέτες μας να σώσουν το ευρώ, δεν περιμένει και ο κόσμος, οι φίλοι μέχρι να αποφασίσουμε εμείς αν θα διαχειριζόμαστε καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τους πόρους. Σήμερα θα πρέπει να αρχίσουμε αυτή την προσπάθεια, όχι αύριο ούτε μεθαύριο. Ευχαριστώ κύριε Γκερπράντη. Σας ευχαριστώ πολύ για την έκθεσή σας. Ολοκληρώνεται έτσι η συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο το μεσημέρι στις 12. Και ερχόμαστε τώρα στο επόμενο σημείο της μέσης διάταξης.